I Θα μιλήσω ισπανικά, λέει ο πρόεδρο, κύριο Κόουσο. Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Μιχαήλ Γιανελίτστε, Υπουργό Εξωτερικών ε, τη Γεωργία. Επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια εβδομάδα μετά την ψηφοφορία που είχαμε εμείς στην Επιτροπή για τις συστάσεις ε, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχέση με την Ανατολική Εταιρική Σχέση. Πριν από την Σύνοδο του Νοεμβρίου του 2017 είναι ένας από τους εταίρους μας η Γεωργία στις ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση που πάντα αναζητεί τρόπους διεύρυνσης των σχέσεών της με την Γεωργία και τη συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ε, συνεργασίας μας. Ε, δεν, σας, ε, δεν θα άλλο, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, με τιμά και με ευχαριστεί ιδιαίτερα η δυνατότητα που βρίσκομαι εδώ ε, να μιλήσω ενώπιον σε φίλους της Γεωργίας για την κοινή μας ιστορία και το κοινό μας μέλλον. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται. Η πρόσφατη έκθεση για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία εγκρίθηκε στην Επιτροπή σας με μεγάλη πλειοψηφία, είναι ακόμα μία απόδειξη της δέσμευσής σας ε, και της προσήλωσής σας προς ε, την ε, Ανατολική Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα του νησηγητή και συνεισηγητέ για την έκθεση περί Ανατολική Εταιρική Σχέση που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα το όραμα. Οι πρωτοβουλίε που εκφράζονται στο έγγραφο που εκπονήσατε και υποστηρίξατε είναι ακριβώ αυτό που ζητεί και έχει ανάγκη σήμερα η Ανατολική Εταιρική Σχέση και ελπίζω να ενισχυθεί για τα επόμενα χρόνια. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας συγχαρώ για την 60η επέτειο από την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά έχουν επιτευχθεί στην περίοδο αυτή, ιδίω ειρήνη, σταθερότητα. Αυτό ξεκίνησε από τη Δύση, ξαπλώθηκε στο κέντρο και στην Ανατολή. Σήμερα είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχει και τόσο ε, πιο πίσω, 27 χρόνια μόλις πριν, ήταν ε, διχασμένη Γερμανία. Η Ενωμένη Γερμανία, η Ενωμένη Ευρώπη είναι ε, πραγματικά μια ελπίδα σε κάποια άλλα μέρη ακόμη του κόσμου. Θέλω να πω ότι η χώρα μου είναι ενθουσιώδης υποστήρικτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλο ποσοστό υποστηρίζουν, των πολιτών μας υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Θέλουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη τα τελευταία δύο δεκαετίες είχαμε αταλάντευτη προσήλωση στα ευρωπαϊκά ιδεώδη και έχουν υποστηριχθεί ε, οι νέοι δημοκρατικοί θεσμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε διέλθει έναν, ε, ευρωπαϊκό, έναν δημοκρατικό μετασχηματισμό ακριβώς λόγω των προσδοκιών που έχουμε να είμαστε πιο στενά συνδεδεμένοι με την Ευρώπη. Και τα τελευταία τρία χρόνια συγκεκριμένα ολοκληρώσαμε τις πιο πολλές από τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στην εταιρική σχέση. έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την ε, πιο ε, εμβαθυμένη αυτή ε, κοινότητα ελεύθερων συναλλαγών. Η ολοκλήρωση συνεχίζεται και κάνει τη θετική διαφορά σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι απλά στόχος εξωτερικής πολιτικής. Είναι και προτεραιότητα στην εγχώρια πολιτική. Ολοκληρώσαμε το θεματολόγιο της πρώτης εταιρική σχέση και έχουμε κατάληξη συμφωνία για το δεύτερο θεματολόγιο, που είναι πιο απαιτητικό και πιο φιλόδοξο, διότι το εκπονήσαμε για πρώτη φορά μαζί με την κοινωνία των πολιτών. Έχουμε επίση ένα νέο σύνταγμα το οποίο πονήθηκε μέσω μιας ανοιχτής διαφανούς διαδικασίας με τη συνεργασία μας με την, ε, σύμβαση, της, ε, την Επιτροπή της Σύμβασης ε, της Γενέβης που καταλήγει ότι με τις πρόοδους αυτές γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την παγίωση και βελτίωση του συνταγματικής τάξης της χώρας με βάση τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η δημοκρατία στη Γεωργία είναι πιο ισχυρή. Από το 2012 είχαμε μεγάλες εξελίξεις. Ανεβήκαμε 37 θέσεις στη διεθνή ε, κατάταξη σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και 28 σε ό,τι αφορά ε, ε, την ελευθερία έκφρασης. Είμαστε πολύ καλύτερα 38 θέσεις ανεβήκαμε σε σχέση με τη διαφθορά. Ε, και έχουμε ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης ε, με βάση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Και είμαστε και πρόεδροι μιας άλλης οργάνωσης ε, πολύ σημαντικής. Is foundation... Ανθρώπινα δικαιώματα είναι το θεμέλιο όλων των μεταρρυθμίσεων που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Υπάρχει στρατηγική για ανθρώπινα δικαιώματα. Νόμος κατά της ακριτικής μεταχείρισης και κατά της ε, βίας σε βάρος των γυναικών. Και αυτά είναι θετικά βήματα. Στη εσωτερική αγορά συμμετέχουμε ως τον δυνατόν περισσότερο. Στο τομέα της τυποποίησης, πιστοποίησης, υγειονομικά, φυτογειονομικά μέσα δικαιώματα πνευματική ειδεξία, ανταγωνισμό, τελωνία, Εμπορικέ σχέσεις. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγαλύτερος εμπορικό εταίρος. αυξάνεται οι εμπορικέ μας συναλλαγέ, αυξάνονται οι εξαγωγές με όλα αυτά τα μέτρα. Καθώς και με τις οικονομικέ μα μεταρρυθμίσεις που δρομολογήσαμε πέρυσι, για να προωθήσουμε την οικονομική μεγέθυνση, νομίζω ότι τα αποτελέσματά μας είναι πολύ θετικά. Με πρόσφατη εκτίμηση του Προέδρου της BRD, η Γεωργία θα είναι ηγέτης ε, ε, στο δεύτερο, στο δεύτερη μέτρων, ε, χωρών συγγνώμη, που προχωρούν τις μεταρρυθμίσεις τους για να προσεγγίσουν τις δυτικές οικονομίες. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων άνοιξε στο, στην Τυφλίδα νέο ε, κατάστημα, ένα γραφείο, εκπροσώπηση εκεί και επενδύει με εκατοντάδες εκατομμύρια. Το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα έχει ξεκινήσει, η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί πρόθεσμα Και έτσι θα προωθηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, η παραγωγικότητα, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα στις εξαγωγές. Αυτά τα λέει και το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε να προωθήσουμε τι δημόσιες επενδύσει για να βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θέλουμε να ρυθμίσουμε την εκπαίδευση, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτή είναι η στόχη μα για το μέλλον. Και οι οίκοι αξιολόγηση παρατηρούν πολύ θετικά. Από το BA3 είμαστε στο BA2 τώρα περάσαμε σίγουρα κάποιους περιφερειακούς κραδασμούς, αλλά ανακάμπτουμε. Και μαζί με την οικονομική ανάπτυξη έχουμε προχωρήσει και στη διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Creative Europe, το ορίζοντα 2020, συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και στο Erasmus Plus. 131 είναι οι χώροι εταίροι, είμαστε στους 10 πρώτους Επίσης συμμετέχουμε στον τομέα των μεταφορών, επικοινωνίων, ενέργειας, ε, ε, γεωργίας, περιβάλλοντος, έρευνας, ε, ανάπτυξης καινοτομία σε προγράμματα. Και στην νότια, αγορά του Νότιου Καυκάσου της ε, συμμετέχουμε στα ανοίγματα της αγοράς και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Επίσης για τον τομέα των οδικών υποδομών και της Βόρειας Θάλασσας, ε, ε, τις λιμενικές ε, υπηρεσίες τις εξελίσσουμε. Προωθούμε και κάποια σχέδια ενεργειακής διέλευσης, διαμετακόμισης, energy, μετάβασης, ενεργειακής μετάβασης. Είμαστε επίσημα σημαντικός εταίρος στο τομέα της ασφάλειας. Φαίνεται αυτό και από την στρατηγική της Ένωση για την ασφάλεια στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση, οργανωμένων εγκλήματο. Επίση, ε, κάνουμε πολλά στι συντηρητικέ απειλέ, καταπολέμηση διακίνηση, ξεγλυνόντο χρήματα. Συμμετέχουμε σε επιχειρήσει διαχείριση κρίσεων, στο Μαλί, για παράδειγμα, στην Κεντρική Αφρική. Και συμμετέχουμε στη σταθερότητα στην Ευρώπη, στι προσπάθειε που αναλαμβάνονται. Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία ξεκίνησαν ένα στρατηγικό διάλογο για θέματα ασφάλειας, για τα θέματα που μας απασχολούν. Όχι μας μόνο, αλλά και την περιοχή και την Ευρώπη. Έχουμε επίσης και πλησιακή στρατηγική συμφωνία συνεργασία με τη Europol και θα ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις και με τη Eurojust. Αγαπητέ κυρίες και κύριοι, έχουμε ε, τη διάσκεψη τον Νοέμβριο. Πάρα πολύ καλή είναι η κατάσταση, ε, έχουμε πετύχει πολλά, πολλά όμω πρέπει να γίνουν ακόμα. και περισσότερα από αυτά που απαιτείται από την Ανατολική Εταιρεία, Γιατί το κάνουμε για εμάς και για το μέλλον της εταιρικής σχέσης, όχι απλά για να κάνουμε το καθήκον ε, όπως προβλέπεται, να κάνουμε τη ε, δουλειά που, και τα μαθήματά μας. Έξι είναι οι βασικοί άξονες που έχουμε μπροστά μας. Πρώτον, όσο το δυνατόν να προσεγγίσει η νομοθεσία μας και οι θεσμικέ πρακτικές μας αυτές τις ένωσης μέσω του θεματολογίου της εταιρικής σχέσης και πέραν. Δεύτερον, ολοκλήρωση με εξειδικευμένου οργανισμού Ένωση για να βελτιωθεί η θεσμική μα ικανότητα και ε, να εκμεταλλευτούμε τεχνογνωσία των Ευρωπαίων συναδέλφων ώστε να έχουμε μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα. Τρίτον, βελτίωση τη αποτελεσματικότητα τη συμμετοχή τη Γεωργία στα ευρωπαϊκά προγράμματα για περισσότερα ωφέλη, πιο ορατά για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να ενταχθούμε σε οικονομικούς, επιστημονικούς, ε, πολιτιστικούς τομείς. Θέλουμε να έχουμε καλύτερο διάλογο τέταρτον για τη διατύπωση και εφαρμογή τομεακών πολιτικών θα δώσει νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη της γεωργίας πέμπτον εμβάθυνση του διαλόγου στην άμυνα για να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερο συντονισμό με τις ε, αμυντικές δομές και δομές ασφάλειας με αμοιβαίο στόχο, με κοινό στόχο τη μεγαλύτερη ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη και στον κόσμο. όπω προείπα πρόσφατα, ξεκίνησε αυτό ο διάλογο. και περιμένουμε να έχουμε πρακτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έκτον, μαζί με την πολιτική και θεσμική ολοκλήρωση θέλουμε μια πιο βαθύτερη ολοκλήρωση στο πέσο τη εσωτερικής αγορά, Δηλαδή σε τομεί όπω μεταφορέ ενέργεια και επικοινωνίες. Όλα αυτά τα project εντάσσονται στις προσπάθειές μας για αποτελεσματική διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε να επενδύσουμε περισσότερο. Να μπούμε στα διαευρωπαϊκά δίκτυα. για να αποδώσουν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς. Όπως βλέπετε, είναι ταυτισμένα τα συμφέροντα Ευρωπαϊκή Ένωση και Γεωργίας. Είναι κοινέ οι αξίες και οι αρχές που μας διέπουν. Και γι' αυτό προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη, βαθύτερη ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε νέα όθηση για να αναζητήσουμε νέες ευκαιρίε, Να προετοιμάσουμε το έδαφος για να επιτύχουμε αυτό το όραμα. Εν ώψη της διάσκεψη ε, του Νοεμβρίου έχουμε τέσσερι προτεραιότητε πιστεύουμε πρέπει να εξεταστούν. Πρώτο, αν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τι φιλοδοξίε και επιλογέ των ενδιαφερομένων μερών και να μείνουν ανοιχτέ οι πόρτε τη. Δεύτερο, ανάπτυξη νέων μέσων χρηματοδοτική βοήθεια και παροχή βοήθεια για να στηριχθούν οι φιλόδοξε μεταρρυθμίσει των συνδεδεμένων εταίρων. Ένα εργαλείο πολύ σημαντικό είναι μεγαλύτερη μόχλευση για την εφαρμογή των προγραμμάτων. Τρίτον, συνδέσεις για παροχή περισσότερων επιχειρηματικών, εμπορικών δραστηριοτήτων. Και οι κοινωνίες πρέπει να έχουν πιο κοντά, με βάση τις κοινέ αξίες. Έχουμε ξεκινήσει ε, τις εργασίες για ανέγερση ενός ευρωπαϊκού σχολείου στη Τυφλίδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επιτρόπο Χάν. Και τέλος, συνεχιζόμενη υποστήριξη στην εδαφική κυριότητα εντός διεθνώς αναγνωσιμένων συνόρων. Είναι σημαντικό ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο τη ειρηνική επίλυση συγκρούσεων. Ξέρετε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ότι υπάρχουν περιοχές της Γεωργίας που είναι υποκατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Νότια Οσετία, Πραγματοσχάρια και Απχαζία. Έχει συνάψει υποτιθέμενε συνθήκες προσχώρησης με αυτές τις περιοχές. Επίσης, έχουμε στην περιοχή Σχοινουάλη ένα παράνομο δημοψήφισμα επίσης εντείνει στρατιωτική της παρουσία στις δύο αυτές περιοχές. Και αυτό απειλεί και την ε, ακαιρεότητα της Γεωργίας αλλά και όλες τις περιοχές. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Απλά να σας πω ότι περισσότερες στρατιωτικές βάσεις έχουν στρατιωτικά συστήματα πολύ προηγμένα, ενώ φιλοξενούν χιλιάδες στρατιώτες και λοιπό προσωπικό. Έχουμε δει ασκήσεις επίσης των ε, ρωσικών ε, ενόπλων δυνάμεων ε, στις κατεχόμενες αυτές περιοχές. Η Ομοσπονδία, η Ρωσική λοιπόν παραγνωρίζει τη δέσμευσή της για μη χρήση βίας. Όπως προβλέπει η παράγραφος 5 της Συμφωνίας Εκεχηρίας του Αυγούστου. Η στρατιωτική παρουσία των Ρώσων στις κατεχόμενες περιοχές δείχνει ότι οι διεθνείς συμφωνίες ε, που έχουν υπογραφεί επιτόπου χρειάζονται διεθνή κάλυψη. Απαιτείται επίσης να ρυθμιστεί το θέμα των σημείων περάσματος ανάμεσα στα διάφορα εδάφη. Η στρατιωτικοποίηση των περιοχών έχει οδηγήσει σε αύξηση της εγκληματικότητας και σε παράνομες απαγωγές Υπάρχει η περίπτωση του χωριού Ρέντβι όπου έχει υπάρξει ουσιαστικά εθνοκάθαρση από πλευράς των Ρώσων και γεωργιανές περιουσίες έχουν σκόπιμα ε, καταστραφή και καεί στα πλαίσια επενδυτικών δίθεν ρωσικών προγραμμάτων είναι βήματα για την περαιτέρω ρωσοποίηση της περιοχής και την προσάρτηση περαιτέρω περιοχών. Οι Γεωργιανοί στην Απχαζία πλέον καταγράφονται ως ξένοι στην ίδια τους την πατρίδα. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αναγκάζονται να ανάξουν επίσης και τα ονόματά τους, τα επίθετά τους, γιατί αλλιώς ε, δυστυχώς δεν έχουν την δυνατότητα ε, φροντίδας στα πλαίσια των δημοσίων συστημάτων υγείας κτλ. Δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στη μητρική του γλώσσα, Η εθνοκάθαρση δυστυχώς συνεχίζεται και οι άνθρωποι που έχουν εκδιωχθεί δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Είναι τμήμα της ε, διαδικασίας ρωσοποίησης και άρνησης της ταυτότητας της Γεωργιανής. Η Επιτροπή Παρατήρησης δεν έχει δυνατότητα πρόσβαση στα κατεχόμενα εδάφη και έτσι δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της. Θέλω όμως να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αποστείλει τους παρατηρητές της η ρωσική κυβέρνηση δυστυχώς ακολουθεί μια πρακτική απαράδεκτη ε, με τρόπους οι οποίοι δεν είναι οι δικοί μας. Εμείς προσπαθούμε με διπλωματικό τρόπο να βρούμε λύση. Η κυβέρνηση της Γεωργίας ε, ε, επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεσμεύεται για την μη χρήση βίας. Εμείς ε, είμαστε πάντα σε επίπεδο διπλωματικής επαφής και συμφιλίωσης και επίσης προσπαθούμε τα ωφέλη από τις επαφές της Γεωργίας με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση να ωφελήσουν και τους κατοίκους της άλλης πλευράς. πρακτικές όπως η υπογραφή της Συμφωνίας Κατάπασης του Πυρός του 2008 δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι η κατοχή εδαφών της Γεωργίας είναι απαράδεκτη ακόμα και σήμερα και χαίρομαι που ασχολείστε με το συγκεκριμένο θέμα στην έκθεσή σας και ευχαριστώ που μάχεστε ακόμα για την ανάκτηση της αδαφικής ακαιρεότητας της χώρας μου. Αγαπητοί φίλοι, θα τελειώσω επαναλαμβάνοντας ότι τα επιτεύγματα των χωρών της Ανατολικής Γειτονίας τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Σαν παράδειγμα η απόφαση για τη χορήγηση θεωρήσεων βραχίας παραμονής δεν ήταν κάτι το εύκολο. Μιας και είναι η πρώτη φορά από το Μάρτιο που μπορώ να πάρω το λόγο μπροστά σας, Θέλω να σας μεταφέρω τις, ε, την ευγνωμοσύνη του γεωργιανού λαού για τις δυνατότητες που δίδεται στους επιχειρηματίες, στους φοιτητές, τους καλλιτέχνες κτλ. Θα προσπαθήσουμε με όλους τους πιθανούς μηχανισμούς να ελέγξουμε κάποιες ε, ε, αρνητικές πλευρές αυτής της διαδικασίας εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια ενημέρωσης εξηγώντας τους πολίτες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το ότι συζητάμε σήμερα εδώ Ελπίζω ότι θα διανύσουμε μαζί τα μελλοντικά βήματα στο πλαίσιο των σχέσεών μας. Ευχαριστώ που με ακούσατε, είμαι στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ο κύριος Μαμίκης έχει το λόγο που είναι μέλος της αντιπροσωπείας με τη Γεωργία. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα μιλήσω λετωνικά. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, γνωρίζοντας πόσο εντατικές είναι οι προσπάθειές σας, η εφαρμογή του ε, προγράμματος ε, σύνδεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γεωργία. Το νέο αυτό πρόγραμμα είναι πολύ καλό και συμφωνώ μαζί σας ότι η Γεωργία είναι μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου οι πολίτες έχουν πίστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζουν το ευρωπαϊκό όραμα. Θα έπρεπε να σας ζηλεύουμε κατά μία έννοια. Ε, λυπάμαι μερικές φορές που οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, δεν έχουν ε, την ίδια πίστη στο ευρωπαϊκό ε, όραμα που έχουν οι πολίτες της Γεωργίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς και τον Πρωθυπουργό σας ε, για τα κοινωνικά προγράμματα που έχετε εφαρμόσει πρόσφατα. Αυτά είναι σημαντικά για τη μείωση της ανεργίας και την ε, αύξηση της ευημερία στη χώρα. Επιτρέψτε μου να σας θέσω μια ερώτηση. Ποιος είναι ο ρόλος σας ως χώρα στην περιφέρεια είσαστε μπροστά όχι μόνο ε, μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών, αλλά γενικά των χωρών υπέρ της Ευρώπης ε, στα νότια του Καυκάσου. Τι ρόλο παίζετε λοιπόν ως χώρα και τι θέλετε να πετύχετε στην ευρύτερη περιφέρεια. Το λόγο θα πάρει η κυρία Αντρικίεν, ε, η οποία ασχολείται με τα θέματα τη ηγήτρια για τα θέματα της Ανατολικής Γειτονίας. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Είναι χαρά που σας ε, βλέπω εδώ στην Επιτροπή μας. Καταρχάς ε, θα ήθελα να αναγνωρίσω και να επενέσω τα επιτεύγματα της χώρας σας όσον αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και την προσέγγιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν είναι μόνο στόχος της εξωτερικής πολιτικής ε, της χώρας σας, αλλά είναι προτεραιότητα και στην εσωτερική πολιτική. Έχετε πετύχει πολλά. Παρ' όλα αυτά απομένει ακόμα δουλειά να γίνει. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων της Συμφωνίας Σύνδεσης και ιδιαίτερα για το ECFPA. Θα εκτιμούσα πολύ την απάντησή σας στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρεμπέκα Χάρμς τώρα, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest. Καλημέρα και από μένα. Όπως ε, είπε ο συνάδελφος, είναι πολύ σημαντικό που ε, ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες ε, για να συζητήσουμε τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την Euronest και τη σημαντική διάσκεψη κορφής που θα γίνει το φθινόπωρο εδώ στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό που η Γεωργία, όπως και άλλες συνδεδεμένες χώρες και τα θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν ε, όχι μόνο υπέρ της συμφωνίας σύνδεσης ε, με τις ε, χώρες αυτές, αλλά είναι έτοιμες να προχωρήσουν και πιο πέρα. Πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν οι προσπάθειες αυτές. Δική μας ε, δουλειά τώρα και το φθινόπωρο είναι να εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι αυτές οι συμφωνίες σύνδεσης ε, είναι κομμάτι της στρατηγικής ασφάλειάς μας δεν έχει ε, απλά να κάνει με καλύτερη ή χειρότερη ανάπτυξη στις γειτονικές μας χώρες. Οι συμφωνίες σύνδεσης και η επιτυχής εφαρμογή τους σχετίζεται όχι μόνο με τη σταθερότητα και τον δρόμο προς τη δημοκρατία στην περιφέρεια, είναι και προς συμφέρον της ε, ασφάλειας και σταθερότητας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αναφέρατε και τα πραγματικά προβλήματα που έχετε με ε, την γειτονική σας χώρα. Η στρατηγική, λοιπόν, ε, ε, επιβαρύνεται από αυτές τις παγωμένες συγκρούσεις που δεν είναι και τόσο παγωμένες, ε, δεν έχουν παγώσει τόσο πολύ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μην αποφύγουμε κατά την συζήτηση της Συμφωνίας Σύνδεσης το βάρος, την επιβάρυνση και την ε, κατοχή εδαφών στις γειτονικές μας χώρες. Τούτου λεχθέντος ε, θα ήθελα να πω κάτι που έχω συζητήσει με την πρέσβηρά σας ε, αλλά και με πρέσβεις άλλων γειτονικών χωρών. Έχει να κάνει με τις ε, πολύ προβληματικές εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία και τον αντίκτυπο που έχουν σε χώρες της γειτονίας μας. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα όμως δημοσίως να υπογραμμίσω ότι η Γεωργία όπως και η Ουκρανία και άλλες γειτονικές χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κοινή στρατηγική ώστε να μην μπορεί ο ε, Τούρκος ε, πρόεδρος να συνεχίσει τις στρατηγικές του και εκτός της χώρας του. Έχουν ζητήσει αρκετή το, ζητήσει αρκετή λόγο για δύο λεπτά ο κάθε ομιλητής παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ να φορέσετε τα ακουστικά σας. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ και σας ευχαριστούμε για την πολύ θετική παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ήρθατε εδώ μία εβδομάδα πριν την συνάντηση της Euronest στο Κίεβο. Έχω μία ερώτηση σχετική με τη Euronest. Η Ουκρανία και η Γεωργία είναι πολύ σημαντικά μέλη της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Η σχέση ανάμεσα στην Ουκρανία και στη Γεωργία πώς μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειες του κυρίου Σακασβίλη στο Κίεβο. Έχουμε το Συμβούλιο Βιετχόνα και πώς μπορεί ο κύριος Σακασβίλη να επηρεάσει τις σχέσεις Γεωργίας και Ουκρανίας. πρόεδρος Σακασβίλη καταπολέμησε την ε, διαφθορά στην Γεωργία. Και ε, φρόντισε για την ε, μετάβαση από το σοβιετικό παρελθόν ε, στο ευρωπαϊκό μέλλον. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Uh, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ πέρα και θα ήθελα να επαναλάβω την υποστήριξή μας για την ε, διαδικασία σταθεροποίησης της ε, δημοκρατίας στην χώρα σας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή η σύγκρουση που έχει παγώσει ουσιαστικά είναι μια πολύ δραματική ε, και επώδυνη κατοχή. Ζείτε σε δύσκολη περιοχή. Η συνάδελφός μου Ρεμπέκα Χάρμς έθεσε ερώτηση σχετικά με την Τουρκία. Και ευχήθηκε να μην υποκύψετε στην πίεση, να κλείσετε σχολεία και να απελάσετε Τούρκους που κατοικούν στη Γεωργία κατόπιν αιτήματος του κυρίου Ερντογάν. Πριν λίγο καιρό είχαμε την ε, περίπτωση του Μουκτζάλη, ε, δημοσιογράφου από το Αζερβαϊτζάν ε, που απάχθηκε στη χώρα σας. Τι μπορείτε να μας πείτε σχετικά με τις έρευνες και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε αυτό. Όσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, αναφερθήκατε στις μεταρρυθμίσεις και χαιρόμαστε που προσπαθήσατε να ανταποκριθείτε στις ε, ε, απαιτήσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Ε, για παράδειγμα, έχετε πει ότι από το 2024 και μετά θα καταργηθεί η άμεση εκλογή Προέδρου. Θα εφαρμοστεί αναλογικό εκλογικό σύστημα. Και μία τελική ερώτηση σχετικά με τον δικαστικό τομέα. Ε, ακούστηκαν πολλές επικρίσεις κατά του ε, ε, δικαστή στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τη Γεωργία, διότι θεωρήθηκε ότι δεν έχει τις απαραίτητες, ε, τα απαραίτητα προσόντα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος και φίλος και εταίρος. Στην έκθεση την οποία συνέγραψε η Επιτροπή μας για τη συνάντηση κορυφής με την Ανατολική Γειτονία ζητήσαμε ε, να υπάρξει διαφοροποίηση για αυτούς που επιθυμούν την εφαρμογή της αρχής more for more. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια Ανατολική Γειτονία plus, συν, για τις χώρες οι οποίες φυσικά έχουν υπογράψει και εμπορικές εταιρικές συμφωνίες. Εσείς ε, αν είχατε αυτή την δυνατότητα, ε, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε. Η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία τι χρειάζονται. Και αυτή η βελτιωμένη συνεργασία ανατολικής ε, γειτονίας με τις πιο προχωρημένες χώρες, αν θέλετε, της περιοχής, σε ποιο βαθμό μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα στις τρεις χώρες τις οποίες προείπα. Και αυτό μήπως θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά και τις υπόλοιπες χώρες οι οποίες κάποια στιγμή θα ενταχθούν στην προσπάθεια. Και τώρα για τις δημοτικές εκλογές την Κυριακή. Τι περιμένετε πώς θα πάνε οι δημοκρατικές εξετάσεις τις οποίες καλείστε να δώσετε για μια ακόμη φορά. Σαφόζερ, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε ως ε, φιλοευρωπαίος πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα όμως μιλήσατε με ξύλινη γλώσσα. Εγώ μπαίνω στη θέση σας και σας θέτω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Ας υποθέσουμε ότι σε πέντε χρόνια η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης αλλά σε διαδικασία αποσύνθεσης γιατί δεν έλυσε τα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα άμυνας και τα προβλήματα ασφαλείας μεταξύ άλλων. Η Γεωργία η οποία είναι μια χώρα ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, τη Ρωσία από τη μία και την Ευρώπη από την άλλη. Έκανε τη σωστή επιλογή, μονομερός προσκολλημένη στην ευρωπαϊκή προοπτική. Σε πέντε χρόνια θα είστε στραμμένοι προς μια Ευρώπη που δεν θα υπάρχει πια όπως την ξέρατε. Η κατάστασή σας θα είναι δύσκολη δεν θα έχετε εταίρος στην Δύση, ενώ στην Ανατολή ε, ο εταίρος σας θα είναι πάντα εκεί. Κάτω από τις συνθήκες αυτές λοιπόν πιστεύετε ότι η πολιτική σας είναι σωστή σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων. Κορβιμίκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. μιλήσω πολωνικά. Υπάρχει ακόμη ένα πρόβλημα στη Γεωργία. Γιαζαρία που ήταν αυτόνομη Σοβιτική Δημοκρατία και την κατέστρεψε την αυτονομία της όχι δική σας κυβέρνηση, αλλά κυβέρνηση του Βίλη. Σε ό,τι αφορά την Οσυρία και την Απχαζία, είναι εθνοτικά διαφορετικές από την Γεωργία και τη φοβούνται τη γεωργιανή κυβέρνηση. Η Ατζαρία. Είχε διαφθαρμένη κυβέρνηση. Ακούω όμως τώρα ότι και η Γεωργία είχε διεφθαρμένη κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση Σακιασβίλη. Πολλά μπορεί να πει κανεί λοιπόν για την κυβέρνηση Σακιασβίλη, αλλά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση τη διαφθορά, νομίζω ότι εκεί τουλάχιστον έκανε πολλά καλά. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε εδώ, κύριε Υπουργέ, για μια ακόμη φορά στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι μαζί θα απογοητεύσουμε όσους στοιχημάτιζαν και στοιχηματίζουν στην αποσύνθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μαζί με τη Μόσχα. Δεν θα πετύχουν. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να, έχετε, να σκεφτείτε ότι μπορεί να έχετε μπροστά σας μια τραγική επιλογή, αλλά ότι μπορεί να συνεχίσετε το μονοπάτι προς την Ευρώπη. Θέλω να σας καλωσορίσω και το γενικό προσανατολισμό της χώρας σας. Τα πιο πολλά από όσα ήθελα να πω υπόθηκαν ήδη από προηγούμενους συναδέλφους. Μια συγκεκριμένη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Έχουμε την συμφωνία τη CFTA. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, πού βλέπετε τη μεγαλύτερη δυσκολία στη διοικητική, η αντιμετώπιση των προβλημάτων ή άλλου είδους πολιτικά ίσως εμπόδια υπάρχουν που καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή της συμφωνίας και αν ναι, σε ποιους τομείς. Αναφέρατε το Σύνταγμα. Από ό,τι φαίνεται στον εκλογικό νόμο είναι θετικό αυτό. Έχετε παρετηθεί του αρχικού σχεδίου να υπήρχαν πόνους για το μεγαλύτερο κόμμα στο, ηλεκτρικό, στο εκλογικό σύστημα. Δεν θα ήταν καλή ιδέα και χαίρομαι που έχει διαγραφεί αυτό και το ίδιο φαίνεται να γίνεται και σε άλλες χώρες που έχουν το ίδιο σύστημα. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Έγινε ένα ερώτημα για την Τουρκία. Είναι γειτονική σας χώρα, ιδίως δε είναι η χώρα που σας συνδέει προς νότον με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν σας ανησυχούν οι εξελίξεις που απομακρύνουν την Τουρκία όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Εμάς μας ανησυχεί πολύ η κατάσταση. Εσάς ε, δεν επηρεάζει τη σχέση σας με τη γειτονική αυτή χώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάλερ. Ελπρόεδρος ο κύριος Φρουντζουλίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και να σας ρωτήσω σήμερα οι σχέσεις με τη Ρωσία σε τι κατάσταση βρίσκονται, έχετε συνομιλίες, έχετε διαπραγματεύσει με τη Ρωσία και πώς, ε, τι έχετε να πείτε σε σχέση με τον επικοινωνιακό πόλεμο που έχει κηρύξει εντό αγωγικών η Ρωσία κατά της Γεωργίας. Το 2008 ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε από τη Ρωσία ε, αυτή η μέθοδος των κυβερνοεπιθέσεων κατά των δυνάμεων της Γεωργίας. Επίσης, τι γίνεται με τους πρόσφυγες. Ξακολουθούν πολλοί γεωργοί να μην ε, μπορούν να γυρίσουν στα σπίτια τους στην Απχαζία και στην Νότια Σετία. Αυτά τα θέσατε στις διεθνείς οργανώσεις ως πρόβλημα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον ΟΑΣΕ, το Συμβουλίο της Ευρώπης, στον ΟΗΕ κτλ. κτλ. Τέλος, ένα εξίσου σημαντικό ερώτημα. Κυρίε και κύριοι, για μένα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς οργανισμοί δεν αντέδρασαν στον πόλεμο του 2008, στον πόλεμο της Γεωργίας, όπως αντέδρασαν μετά την ρωσική επίθεση στην Ανατολική Ουκρανία. Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, ε, αλλά ποια είναι η δική σας άποψη. Και πάλι ε, κάτι τελευταίο, προσωπική άποψη. Η Γεωργία πρέπει να γίνει δεχτή ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον πληρεί τα, τις υποχρεώσεις. Με βάση το κυπριακό μοντέλο. Η κυπριακή δημοκρατία έγινε δεκτή ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το βόρειο τμήμα να είναι κατεχόμενο από την Τουρκία. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να γίνει και με τη δημοκρατία της Γεωργίας. Έτσι θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα παράδειγμα ότι δέχεται την Γεωργία ως μέλος Ένωσης με τα κανονικά της στα σύνορη. Τελευταία ομιλείται κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Υπουργέ που ήρθατε εδώ για να κάνετε κάτι που εμείς δεν κάνουμε αρκετά, δηλαδή να εκφράσετε την ικανοποίησή σας και να χαιρετήσετε τα επιτεύγματα των όσων έχει πετύχει η χώρα σας. Η παρουσία σας είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτη μας μιλήσετε για την DCFTA, τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι έχει αντλήσει η χώρα σας από αυτά και είναι ιδιαίτερα ε, θετικά. Ένας από τους λόγους που έχουμε αυτά τα ωφέλη και τα ε, ευεργετήματα, και είναι σαφές ότι μιλήσετε υπέρ τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λόγω του ότι έχετε βάλει το, στο επίκεντρο το λαό σας. Είπατε ότι δεν ε, Καλύπτεται απλά τα καθήκοντα και κάνετε τα μαθήματά σα, αλλά ότι έχετε βάλει στο επίκεντρο τον πολίτη. Αυτό μπορούμε να δούμε και νομίζω ότι το βλέπετε και εσείς από τα σχόλια των συναδέλφων είναι ότι σας στηρίζουμε. Στηρίζουμε και εσάς, το έδατε στο ψήφισμα και φαντάζομαι το έχετε δει και με πολλούς άλλους τρόπους στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαξένωσης Ένωση Γεωργίας. Και ρητίνη και υποστήριξή μας προς την εδαφική σας ακεραιότητα. Να είστε παρακαλώ βέβαιος ως προς αυτό. Επίσης, πολύ σωστά στα σχολιά σας. Μας κάνατε, αναφέρει ένα κατάλογο στιγμάτων που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Θα μας βοηθούσε να ξέρουμε τις δικές σας προτεραιότητες στο πλαίσιο αυτού του καταλόγου. Έρχεται το Euronest και έρχεται και η διάσκεψη εδώ στις Βρυξέλλες. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να βάλουμε στην κορυφή του καταλόγου των προτεραιοτήτων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μούντι. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να απαντήσετε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για το μεγάλο σας ενδιαφέρον για τη Γεωργία. Και σας ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, οι οποίες δείχνουν για άλλη μια φορά την αφοσίωσή σας στην ε, βελτίωση των σχέσεων ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Γεωργίας. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέθηκαν πολύ σημαντικές ερωτήσεις και έχω μόνο 10 λεπτά να απαντήσω. Γι' αυτό θα προσπαθήσω σύντομα να απαντήσω σε όλες. Καταρχάς όσον αφορά το ρόλο της γεωργίας ε, στην ευρύτερη περιφέρεια. Η γεωργία θέλει να δώσει ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή είναι η πολιτική που επιδιώκουμε να εφαρμόσουμε και αυτές είναι οι σχέσεις που θέλουμε να έχουμε με τις χώρες της ε, περιφέρειας. Αυτό είναι που κινεί όλες τις μεταρρυθμίσεις και όλες τις δραστηριότητες της Γεωργίας. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φίλων μας, ε, την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Θέλουμε να είμαστε τμήμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, καθώς και των ευρωπαϊκών οικονομικών ευκαιριών. αναπτύσσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας όχι μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε στενή συνεργασία με χώρες της Κεντρικής Ασίας της ε, από Ανατολής και πιστεύουμε ότι η Γεωργία είναι αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κόμβο ε, στις συναλλαγές ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ασία. Όσον αφορά την Τουρκία αναφέρθηκε αρκετές φορές. Συνεργαζόμαστε μαζί της σε ε, προγράμματα στρατηγικής σημασίας για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι ο αυτοκινητόδρομος ε, που θα συνδέσει με την Τυφλίδα, που θα εγκαινιαστεί στις 30 Οκτωβρίου. Ε, αυτό αποτελεί καρπό εργασιών πολλών χρόνων και συνεργασίας με το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία και έτσι δημιουργείται νέα σύνδεση Ασίας και Ευρώπης. Συνεργαζόμαστε με τις δύο αυτές χώρες και πάνω σε στρατηγικά ε, θέματα όπως είναι η παροχή αερίου στην ε, Ευρώπη και πόρων από την Κασπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη υπάρχουν αγωγοί, ενώ ε, αναπτύσσονται και νέοι. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στρατηγικά προγράμματα τα οποία ε, μας συνδέουν με την Τουρκία και μας ενδιαφέρει να πετύχουν τα προγράμματα αυτά, αυτά τα προγράμματα συνεργασίας. Ελπίζουμε και πιστεύουμε κάποια θέματα επίμαχα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία και θέματα που επηρεάζουν την περιοχή. Ελπίζουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα επιληθούν και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ε, ευρωατλαντική κοινότητα και να έχουμε τέρους προς όλες τις κατευθύνσεις. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να, συνεργασ... να συνεργαζόμαστε όχι μόνο με τις χώρες που ανέφερα, αλλά οικοδομούμε και στενές σχέσεις με συνδεδεμένες χώρες. Ε, αναφέρθηκε το θέμα των σχέσεων ε, με τη Μολδαβία και την ε, Ουκρανία και τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές, αλλά και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών. Έχουμε λοιπόν ε, εις βάθος διάλογο και με τις δύο αυτές χώρες, τη Μολδαβία και την Ουκρανία και εξερευνούμε τις δυνατότητες εξετάζουμε νέα βήματα Ολοκλήρωση Θέλουμε να ε, εκμεταλλευτούμε όλα τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας και να προδρεύσουμε στις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει η επιτυχία και των συνδεδεμένων χωρών ε, και όλων των χωρών όμως ε, της ανατολικής γειτονίας. Η Ανατολική Γειτονία είναι πρόγραμμα μεγάλης σημασίας για όλα τα μέλη της. Πιστεύω ότι το ίδιο πνεύμα δεσπόζει εδώ και θα δεσπόσει και κατά τη διάρκεια της ε, συνάντησης κορυφής. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές όσον αφορά το επίπεδο ε, φιλοδοξίας. Ε, σημαντικό όμως είναι να υπάρχει ενότητα όσον αφορά τις αρχές της ε, ανατολικής γειτονίας. Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε για την επιτυχία αυτού του σημαντικού προγράμματος. Από την άλλη σημαντικό είναι να αφήσουμε και ανοιχτούς τους διμερείς διάβλους στην ε, Ανατολική Γειτονία. Η Γεωργία θα συνεχίσει να ε, συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω την απάντηση της επόμενης ερώτησης. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες. Έχουμε επισημάνει έξι προτεραιότητες στην ε, διμερή διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική μας όμως προτεραιότητα είναι πολιτική και πρόκειται για την υποστήριξη η οποία θα πρέπει να συνεχιστεί όσον αφορά τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και τις ευρωπαϊκές επιλογές της γεωργίας. Αυτό λοιπόν ε, θα αποτελέσει το κίνητρο και για άλλες επιτυχίες στο μέλλον. Όσον αφορά εσωτερικά θέματα, θα ήθελα πρώτα να ολοκληρώσω όσον αφορά τους ε, γειτόνους μας. Ε, τέθηκε ερώτηση σχετικά με την Ουκρανία και την Ουκρανία. Έχουμε πολύ ισχυρούς δεσμούς με την Ουκρανία. Είχαμε πολλές επαφές, είχαμε ε, επίσκεψη του δικού μας Πρωθυπουργού στην Ουκρανία, του Πρόεδρου της Ουκρανίας ε, στη χώρα μας ε, και γενικά έχουμε πολύ στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών που δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες προσωπικότητες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι δεν θα υπάρξουν προσωπικότητες που θα παρέμβουν αρνητικά στις σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών χωρών όσον αφορά τις εσωτερικές υποθέσεις. Καταρχάς το Σύνταγμα. Όπως ανέφερα, το έγγραφο είναι πολύ προοδευτικό, ε, έχει ε, εγκριθεί από την Επιτροπή της Βενετίας και προβλέπει νέα κοινωνικά περιβαλλοντικά δικαιώματα, ελευθερίες ε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, και λοιπά. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της ε, Γεωργίας προβλέπει και τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό έγγραφο για την Γεωργία. Και πιστεύουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια όλα αυτά θα είναι εμφανή για όλους και εσωτερικά στη χώρα και εξωτερικά. Οι αλλαγές αυτές ε, θα διασφαλίσουν ε, πολιτικό πλουραλισμό και δυνατότητες ε, για την αντιπολίτευση. όσον αφορά την κατάργηση του συστήματος ε, των μπόνους Ζητήθηκαν προεδρικές εκλογές ε, με άμεση ψηφοφορία. Οι αλλαγές ε, λοιπόν του νέου εκλογικού συστήματος και για το Κοινοβούλιο και για τον Πρόεδρο. Ε, θα εφαρμοστεί το 2024. Αυτό αποτελεί σημαντικό επίτευγμα της χώρας μας. Όσον αφορά άλλες εκλογές, ε, ναι, βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο. 21 Οκτωβρίου θα έχουμε ε, δημοτικές εκλογές. Έχουμε παρατηρητές από τον ΩΣΑ, καθώς και από άλλους ε, φορείς παρακολούθησης εκλογών. Όλες οι δηλώσεις του δείχνουν ότι έχουμε ελεύθερες και δίκαιες διαδικασίες και είμαι βέβαιος ότι και αυτό θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία της δημοκρατίας μας. Η Γεωργία θέλει να διασφαλίσει δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους πολίτες μας. και η εφαρμογή ευρωπαϊκών ε, προτύπων ε, και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον τρόπο να εισάγουμε τους πολίτες μας σε μια κοινότητα και σε ένα περιβάλλον που θα ωφελήσει όλους τους πολίτες της χώρας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να ε, διαδώσουμε τα ωφέλη της ε, ανάπτυξής μας και του θεματολογίου μας, ε, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες της Γεωργίας συμπεριλαμβανομένων αυτών που ζουν στις κατεχόμενες περιοχές. Ε, έχουμε θίξει θέματα που σχετίζονται με ε, τις κατεχόμενες περιοχές ε, και είχαμε πολύ σημαντικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καθώς και του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων φέτος τον Μάρτιο αναφέρθηκε η ανάγκη προσέλευσης του είπα του αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις κατεχόμενες περιοχές. Ωστόσο δεν δόθηκε η ευκαιρία αυτή. Έχουμε όμως την υποστήριξη των ε, ευρωπαϊκών χωρών στο ψήφισμα αυτό και προσβλέπουμε στη συνέχιση των εργασιών με την υποστήριξή σας ώστε να μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα με βάση αυτά τα διεθνή μέσα. Είχαμε ισχυρότερη υποστήριξη από τα προηγούμενα χρόνια και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε την τακτική έκθεση του Γενικού Γραμματέα καθώς και απόφαση ε, των ε, αναπληρωτών υπουργών που αναφέρονται σε σημαντικές ε, παραβάσεις από πλευράς της Ρωσίας στις κατεχόμενες περιοχές, ε, καθώς ε, και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρώσει η ρωσική πλευρά. Αυτό δεν αρκεί. Εργαζόμαστε όχι μόνο μέσω διεθνών οργανισμών, αλλά και στις ε, συζητήσεις μας ε, γενικότερα και με την υποστήριξη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ελπίζουμε ότι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι θα μπορέσουν να επανέλθουν στις χώρες τους, στους τόπους τους. Λυπάμαι που δεν ε, είχα το χρόνο να απαντήσω σε πολλές από τις ερωτήσεις λόγω του χρονικού περιορισμού. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε ε, τον διάλογο αυτόν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και την ανταλλαγή απόψεων με τους ε, υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Thank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 So, Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 5. Μέχρι τις 11 παρα 10 έχουμε χρόνο πρέπει να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της ΚΕΠΑ. Η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων από πλευράς μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος, ιδιαίτερα τους κοιόδης των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, συμφωνήσαμε σε 24 συμβιβαστικές μετά από αίτημα συναδέλφων αποφάσισα να καταφέσω και κάποιες νέες συμβιβαστικές για την ΚΕΠΑ και έχουμε συμπεριλάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα έκκληση γύρω από την πολιτική αυτή και για τη Μέση Ανατολή και για το Ιράν και υπάρχει και μία παράγραφος για τον προϋπολογισμό και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Νομίζω ότι με τις νέες αυτές προτάσεις το τελικό κείμενο θα θεωρηθεί πλήρες. Μία τελευταία παρατήρηση να θυμίσω σε όλους ότι έχουμε μία έκθεση CSDP και τις περιφερειακές εκθέσεις μπροστά μας και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν θέλω να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας τόσο στις επιμέρους χώρες και περιοχές και υπήρους. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με εγκυκλοπαιδικό τρόπο, αλλά με στρατηγικό, αποδίδοντας την κεπάτη σημασία που έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους για τη βοήθειά τους και θα δώσω το λόγο στους Κιώδης. Ο Φλέκενστάιν δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Εκπροσωπώ τον Κνούτ, εξ ονόματος του λοιπόν και των σοσιαλιστών, να πω ότι είχαμε πράγματι μια πολύ παραγωγική συνάντηση. Οι συμβιβαστικές είναι ισχυρές τροπολογίες, μας καλύπτουν. Υποστηρίζουμε την άποψη να μην είμαστε τόσο συγκεκριμένοι σε επιμέρους χώρες και θέλω να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους Σκιώδης και τον Ντέιβιντ για την πολύ καλή τους δουλειά. Ευχαριστώ καθηπήρη. ο κύριος Πάιτ που αντικαθιστά τον κύριο Βαντάλ. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων θα ήθελα να πω ότι το κείμενο αυτό μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Είναι σαφές, καλύπτονται πολλά δύσκολα θέματα, όπως η ατυχής περίπτωση των βίαιων στρατιωτικών ενεργειών των Ρώσων στην Ουκρανία, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το θέμα της μετανάστευσης κτλ. Κάποια συγκεκριμένα θέματα αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο, η ανάγκη για περαιτέρω αμυντική συνεργασία είναι καιρός να την βελτιώσουμε, να την αυξήσουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι σημαντικό είναι οι βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνασφάλειας, είναι κάτι που ανήκει όλο και περισσότερο στην κοινή εξωτερική πολιτική και ασφάλεια σε συνεργασία βέβαια με τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ λοιπόν και τον εισηγητή και τους Σκιώδης και φυσικά θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή. Η κυρία Λούσινγκ από την QNGL. Ευχαριστώ πολύ. αν και είναι πολύ πρακτική η προσέγγιση του εισηγητή και η πολιτική άμυνας και ασφαλείας, η εξωτερική πολιτική είναι το θέμα, θεωρούμε προβληματικό το ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη ότι οι περισσότερες αιτίες συγκρούσεων είναι κοινωνικής φύσης και αποτελούν ε, αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος, ε, περιβαλλοντικών προβλημάτων κλπ. Η, πρόταση, η, η έκθεση θεωρεί ότι και αυτού του τύπου τα προβλήματα θα πρέπει να λυθούν ε, στρατιωτικά. Δεν έχουν υιοθετηθεί οι τροπολογίες μας, ε, ωστόσο θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποια καλά στοιχεία στο σχέδιο έκθεσης, ε, ιδιαίτερα τις συμβεστικές προτάσεις 8 και 27 στηρίζουμε, δεν θα σας τις ε, διαβάσω. Όσον αφορά άλλες συμβαστικές προτάσεις, Ε, δεν ε, είναι συμβατές ε, με την βασική μας θέση και αναφέρομαι ιδιαίτερα στις συμβαστικές τροπολογίες που λαμβάνουν υπόψη τις τροπολογίες ακροδεξιών κομμάτων. Αυτό λοιπόν ε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα υποβάλουμε ε, ε, έκθεση της μειοψηφίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λουέζινγκ, για τα λόγια σας. το περίμενα και αυτό. Ο κύριος Σαφοζέρ, παρακαλώ. Ναι, μπορείτε να το προφέρετε και στα γερμανικά το όνομά μου, γιατί είναι γερμανικής προέλευσης. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και δεν υποστηρίζουμε αυτό το κείμενο, πάντως, αν με επιτρέπετε, ένα μικρό ιντερλούδιο για τη γαλλογερμανική συζήτηση. Ο πρόεδρος μας λέει θα το ε, υποστήριξει αυτό το κείμενο, διότι μιλάει για την ευρωπαϊκή κυριαρχία. Εγώ δεν συμφωνώ. ενώ κάπως απαρνείται της εθνική, την εθνική διάσταση εμέσως. Πρέπει όμως να είμαστε συνεπείς, να πούμε ότι χρειάζεται ένας προϋπολογισμός για την Ευρωζώνη ή ένας ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Η Γερμανία όμως δεν δίνει την σύμφωνη γνώμη της προς το πάνω για κάτι τέτοιο. Τι θέλουμε λοιπόν. Ή όπως εμείς είμαστε κατά της ευρωπαϊκής κυριαρχίας γιατί προστηρίζουμε την εθνική διάσταση ή ακολουθούμε μια άλλη λογική, τη δική σας, μια ευρωπαϊκή λογική, όμως τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί ευρωπαϊκό προπολογισμό. Δεν μπορούμε και να λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά και να αρνούμαστε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαφχάουζερ. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Η CR πράσινη, η FTD, όχι. Επομένως, να σας αναφέρω για μια φορά το χρονοδιάγραμμα. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιήσει στην Επιτροπή Εξωτερικών στις 6 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις και μπορούμε να περάσουμε ήδη στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. 15 λεπτά νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Σύστασε προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΕ σχετικά με το Χονγκ Κόνγκ 20 χρόνια μετά την παράδοσή του. Να ξαναδώσω στον κύριο Κόουσο την Προεδρία παρακαλώ. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 6 για τη σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΙΕΔ σε σχέση με το Hong Kong 20 χρόνια μετά την παράδοσή του. Είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά εμπορικά κέντρα το Hong Kong ακόμη και σήμερα υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή τον Άλεν Σμιθ για να μας παρουσιάσει το σχέδιο ε, έκθεσης που κατέθεσε πριν από τρεις εβδομάδες. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Σα παρουσιάσω τι δικέ μου συστάσει. Ευρύ το φάσμα που καλύψαμε. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό και τη γραμματεία γιατί εργάστηκαν σκληρά και το δικό μου συνεργάτη. Συναντήσαμε διάφορους εμπλεκομένους φορές, την αποστολή της Κίνας και του Χονγκ Κόνγκ, στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Αποστολή στο Χονγκ Κόνγκ και γενικώ όλοι είχαν μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση. Η προσέγγιση μας ήταν να παραμείνουμε στα πραγματικά γεγονότα. Ε, είναι σημαντικό εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συλλογικά να βελτιστοποιήσει και να μην γιστοποιήσει την εθνική συνεισφορά και να έχουμε μια έκθεση που θα μιλά για αξίε και για την πραγματική κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, που φυσικά είναι πολύ σημαντικό μέρος, ε, κομμάτι μιας χώρας πολύ σημαντικής ε, για την Ένωση. Δεν θέλαμε να ήμασταν κριτικοί, επικριτικοί και να δείχνουμε το δάχτυλο, ιδίω γιατί έχουμε να μάθουμε πολλά σε ό,τι αποβλήτων ε, και την ενεργειακή απόδοση και βέβαια και υπάρχουν τα συστήματα δημοκρατίας, ε, δικαστική, ε, δικαστικό σύστημα, μια χώρα δύο συστήματα. Ε, περιμένω βέβαια να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και είμαι πολύ ανοιχτός και στην κατάσταση τροπολογιών γιατί θέλω να έχουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση στην Επιτροπή μας για την έκθεση αυτή. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας σχόλια. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους και όσους ε, Η πρώτη είναι η κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για αυτό το σχέδιο έκθεσης, αλλά και τους ανθρώπους από τη Γραμματεία και, από το, και τους συνεργάτες μου που με βοήθησαν. Όπως γνωρίζετε, είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Έχουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 24 Οκτωβρίου και θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την έκθεσή σας. Ε, γνωρίζετε ότι το Χονγκ Κόνγκ είναι πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος για την Ευρώπη και είναι σημαντική και η κατάσταση της δημοκρατίας εκεί. Μία χώρα, δύο συστήματα είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και αυτό εξηγεί γιατί το Χονγκ Κονγκ είναι 15ο ε, στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπροστά από πολλές, ε, πολύ μεγαλύτερες χώρες. Όπως γνωρίζετε, το Χονγκ Κονγκ έχει αυξήσει τη συνεργασία με το πρόγραμμα Εράσμους στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και με άλλα προγράμματα κινητικότητας. Και συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Περιμένω λοιπόν ε, να δω τροποποιημένο το σχέδιο έκθεσης. Και σας ευχαριστώ πολύ για την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λάινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μιλώ εκ μέρους ε, του κυρίου Πίκουλα, σκιώδους εισηγητή μας, ε, που ζητεί συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά το θέμα της εκείνας με ενδιαφέρει και εμένα πολύ. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή λοιπόν αποτελεί μια καλή επισκόπηση της κατάστασης στο Χονγκ Κόνγκ 20 χρόνια μετά την παράδοση. Δεν έχουμε δώσει πολύ σημασία στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια. Είχαμε δύο ψηφίσματα για τους ε, βιβλιοπόλες που εξαφανίστηκαν, αλλά γενικά ε, ήμασταν αρκετά σιωπηλοί στο θέμα αυτό, γι' αυτό νομίζω ότι η έκθεση αυτή εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή. Μην σας πω ότι καθυστέρησε κιόλας. Ε, το επίκεντρό μας θα πρέπει να είναι το μία χώρα, δύο συστήματα. Αυτό το είχαν υποσχεθεί για 50 χρόνια. Τα 20 χρόνια τώρα ήδη πέρασαν, άλλα 30 χρόνια απομένουν. Και θα μπορούσε κανείς να κάνει διάφορες παρατηρήσεις σχετικά με το καθεστώς αυτό. Είδαμε με διάφορες παρεμβάσεις του Πεκίνου με διάφορες επεμβάσεις του Πεκίνου στην ε, πολιτική του Χονγκ Κονγκ ότι πολλοί δημοσιογράφοι δεν γράφουν πια αυτά που ήθελαν να γράφουν. Είδαμε τους βιβλιοπόλες Αυτά λοιπόν είναι γεγονότα που ε, ε, αντιφάσκουν με το ε, μία χώρα δύο συστήματα. Βέβαια ήταν και εκτενείς οι διαμαρτυρίες στο Χονγκ Κονγκ. Υπάρχουν πολλοί που θέλουν όχι μόνο μία χώρα δύο συστήματα, θέλουν και την ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ. Ε, οι παρατηρήσεις μας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και αυτά. Ε, ο εισηγητής ε, εξετάζει τα προβλήματα του Χονγκ Κονγκ που είναι τα προβλήματα μιας μεγάλης πόλης, 10 εκατομμύρια, η διαχείριση των απορριμμάτων, ε, μετανάστευση, όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά κάνει να έχει στενή σχέση με το Χονγκ και ε, πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή θα περιγράψει το επόμενο στάδιο σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Χονγκ Κονγκ. Προσβλέπω στη συνέχεια των εργασιών. Ο κύριος Μπέλτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σμιθ, διάβασα με μεγάλη χαρά την έκθεσή σας. Ιδίω μετά τα όσα διαβάσαμε στον τύπο τις τελευταίες μέρες για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ. υπάρχει το θέμα της ε, στάσης τους απέναντι ε, στην λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Διάβασα και ξαναδιάβασα το κείμενό σας. Και από ό,τι βλέπω, περιγράφεται με πολύ πλήρη τρόπο την κατάσταση, γι' αυτό πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια. Και μεταφέρατε πιστά την πραγματικότητα. Αν μου επιτρέπετε, λείπει μία παρατήρηση στις συστάσεις. Μιλάτε μεν για αυτή την κατάσταση μια χώρα δύο συστήματα. Νομίζω όμως ότι όπως είπε και ο συνάδελφος Γιολάινου πρέπει να εστιάσουμε στα γεγονότα. Να δούμε τι έγινε και με αυτούς ε, τους εκδότες και καλό θα ήταν σε ό,τι αφορά την ισορροπία να είστε λίγο πιο προσεκτικός σε αυτή την παράγραφο. να τροποποιήσετε ίσως ε, την παράγραφο αυτή. Για να είναι σωστά και, σωστή και η μεταφορά των γεγονότων ε, και η ερμηνεία. Θα τα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες για να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ο κύριος Σπάιτ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ότι είναι πολύ καλή η έκθεση. Είναι μια ανοιχτή άθουσα κοινωνία, κοινωνία του Χονγκ και πρέπει να υποστηρίξουμε τη συνέχιση των προοπτικών αυτών. Έχουμε την αρχή μια χώρα δύο συστήματα που είναι πολύ βασική για το σκοπό αυτό. Υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προβληματικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν παρενόχληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των υποστηρικτών της δημοκρατίας, υποβάθμιση της ελευθεροτυπίας, ενίσχυση των ελέγχων σε ό,τι αφορά την πώληση ευαίσθητων ποτικών βιβλίων. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο, Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το ζήτημα της ξεπλήματο χρήματος βορειοκορεατικού χρήματος στο Χονγκ Αυτό παραβιάζει τη, το ψήφισμα του, του Συμβουλίου Ασφαλείας που μιλάει για να μην, την απαγόρευση κοινοπραξιών με τη Βόρεια Κόρη. ευχαριστώ. Ξαναδώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Σμιθ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι μου ενθάρρυναν τα ε, σχόλιά σας. Νομίζω ότι θέλετε ένα πιο, ε, μια πιο ισχυρή διατύπωση και ελπίζω να έχω τις τρόπολογές σας για τους οικονομικούς δεσμούς, ε, τη διακυβέρνηση, την εργασία. Και καλά λέτε και χαίρομαι που το λέτε ότι είναι καλό να δούμε μετά την 25 από την παράδοση τι γίνεται στο Χονκό και να το ακολουθούμε με επικοδομητικό πνεύμα. Θα μιλήσω για τη δικαστική ανεξαρτησία και την το τύπο με πιο ε, ισχυρές διατυπώσεις. Πράγματι υπάρχουν κάποιοι φορείς στο Χονγκ που αναζητούν που ζητούν μάλλον την ανεξαρτησία του Χονκό Θα πρέπει όμως να δούμε ε, γίνεται, την κυρίαρχη θέση του Χονγκ δεν την αμφισβητούμε και στο έγγραφο μας προσπαθούμε να δούμε και τι συζήτηση γίνεται εντός του Χονγκ αλλά και το ποια είναι η πραγματικότητα που νομίζω ότι είναι ακριβώς εκεί που έπρεπε να είμαστε. Θα προσπαθήσω για το Τζέι που λέτε την παράγραφο αυτή να έχω μια διατύπωση καλύτερη και θα περιμένω και τις τροπολογίες σας για να περιληφθεί μια αναφορά στην Κορέα και στο ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε μιλήσει για διάλογο με την Ταϊβάν και αλλού. Εντάξει, το Χονγκ Κόνγκ δεν είναι μια μονομένη περίπτωση. Νομίζω πρέπει να δούμε την ευρύτερη κατάσταση για το ξέπλυμα χρήματος που είναι μια μείζων ανησυχία και σε σχέση με το Χονγκ Κόνγκ. Κάποια χρόνια πριν είχα πάει εκεί και ήταν τότε πρόβλημα το ξέπλυμα χρήματος όπως είναι και σήμερα. Προσπάθειες έχουν γίνει αλλά μπορούν να γίνουν περισσότερες ε, κοινέ προσπάθειες. Περιμένω λοιπόν τις ε, τροπολογία σας ελπίζοντας να φτάσουμε σε μια ως το μεγαλύτερη συνένεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 24 Οκτωβρίου. Κανονικά θα έχουμε μια δεύτερη συνεδρίαση στις 20 ε, Νοεμβρίου. Το επόμενο θέμα γίνεται μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Θα διακόψουμε μέχρι τις 11. 10 minutes. AUTHORWAVE colleagues, the last point. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήρθαμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής ε, ημερήσιας διάταξης που είναι η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Θα το συζητήσουμε από κοινού με την ε, Επιτροπή Ανάπτυξη. Θέλω να καλωσορίσω του συζητητέ μα ε, από τα θεσμικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον Κουν Φερβέκ, εκτελεστικό διευθυντή για την Αφρική, συγγνώμη, από την ΕΙΕΔ. Έχουμε την κυρία Κάρλα Μοντέση, διευθύντρια για τη Κεντρική Αφρική στην Γενική Διευθυνσή ΔΕΦΚΟ, την κυρία Σουζάνε Μαλάουν, προϊσταμένη μονάδα για τη Βόρεια Δυτική Κεντρική Αφρική στο ΕΚΟ. Θέλω να καλωσορίσω και την κυρία Νατζάτ Ρότζι, αναπληρωτή ειδική εντεταλμένη για την πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή σταθεροποίηση της κεντροαφρικανική Δημοκρατίας. Ε, θα έχουμε λοιπόν σε δύο μέρη την ανταλλαγή απόψεων. Καταρχάς, θα ακούσουμε γενικά πώς βλέπει τα πάντα Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ακούσουμε του εκπροσώπους τη ΕΕ και τη ε, Κομισιόν και θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος ερωταπαντήσεων και μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ε, την ε, αναπληρώτερη ειδική εντεταλμένη για την Μινούσκα. Είναι σημαντικές οι προκλήσεις ε, στο, ε, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το είπε και ο πρόεδρος Κεντροαφρικανικής ε, Δημοκρατίας. Από το 2017 έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της ασφάλειας. Έχουμε βία από ενόπλες ομάδες με πολλά θύματα και μεταξύ του άμαχου πληθυσμού πάνω απ' όλα η χώρα χρειάζεται τη διεθνή βοήθεια. Γι' αυτό λοιπόν ε, πιστεύω πολύ επίκαιρη η σημερινή συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Από όλε τι πτυχέ θα πιάσουμε το θέμα, την πολιτική κατάσταση, την ασφάλεια, την ανάπτυξη, την ανθρωπιστική βοήθεια. Πριν δώσω το λόγο στου ομιλητέ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ντεβε, το Στέλιο Κούλογλου, για να μα κάνει και αυτό μια εισαγωγική τοποθέτηση. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που πήρε την πρωτοβουλία να ενημερώσει τα μέλη των Επιτροπών μας για την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. What we need to do now is not uh, just uh, speaking about this δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για αυτή τη χώρα βέβαια. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες απαντήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον της χώρας αυτής. Μέχρι το 2014 η κεντροαφρικανική δημοκρατία ε, ήταν ορφανή διεθνούς βοήθειας, έπαιρνε μόνο, δεχόταν μόνο μια πολύ μικρή στήριξη από τις ε, ε, από τις κοινότητες χωρών που δίδουν ε, βοήθεια, αν και είναι από τις πιο φτωχές χώρες λόγω απεικιοκρατίας, συγκρούσεων, εμφυλίων συγκρούσεων, στρατιωτικών πραξικοπημάτων, ε, επιθετικών καταστρεπτικών για τη χώρα ελίτ και ιδιαίτερα εύθραστων και ευάλωτων θεσμών. Από το 2013 όμως ε, υπήρξε εκτοπισμός ε, ενός εκατομμυρίου κατοίκων της περιοχής αυτής, το 20% δηλαδή του πληθυσμού και αυτό ολοκληρώθηκε το 2014. Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να επανεμπλακούν αποκαθιστώντας την ειρήνη και βελτιώνοντας τις προοπτικές. Τον Ιούλιο του 2014 η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησαν ένα καταπίστευμα με ένα αρχικό προϋπολογισμό 64 εκατομμυρίων που αυξήθηκε στα 230 εκατομμύρια και από αυτό ε, είναι αδιάφετα τα 110. Ε, βέβαια τα μέσα ενημέρωσης, τα κυρίαρχα τουλάχιστον, σκοτίστηκαν για την κατάσταση στην Αφρικανική. Αλλά η κατάσταση φαίνεται ότι δεν έχει βελτιωθεί. μετά από τις πρώτες διεθνείς πρωτοβουλίες. Υπάρχουν κάποια σχετικά καλά νέα. Τον Ιούλιο ε, στα πλαίσια του νέου οδικού χάρτη ε, για τη συμφιλίωση υπό την αιγίδα της, του Οργανισμού Αφρικανικής Ενότητας, αλλά δυστυχώς η βία συνεχίζεται. Η κατάσταση σε επίπεδο ασφαλείας είναι πραγματικά ανησυχητική, όπως ε, παρατηρείται και σε μια πρόσφατη έκθεση του International Crisis Group και του Human Rights Watch. Ε, δολοφονίες αμάχων, σεξουαλική βία, εμπλοκή μάλιστα και παιδιών σε αυτές τις απαράδεκτες καταστάσεις ε, και δυστυχώς τα πράγματα τείνουν να ξεφεύγουν από κάθε μορφή ελέγχου. Τον Ιούνιο για πρώτη φορά ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων ξεπέρασε τους 500.000 και άλλοι τόσοι περίπου ε, ζουν σε γειτονικές χώρες ε, ως πρόσφυγες. Όλοι γνωρίζουμε ε, ότι η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς, οι δυσκολίες είναι τεράστιες και γι' αυτό σήμερα καλούμεθα να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα πολύ σημαντικά. Πώς, σαν παράδειγμα, να μετατρέψουμε τις κρατικές δομές σαν κάτι το οποίο οι πολίτες θα θεωρήσουν προστατευτικό και υποστηρικτικό για αυτούς. Δεύτερον, πώς ε, να τροποποιήσουμε μια οικονομία που βασίζεται στις συγκρούσεις, τους εκβιασμούς, τις καταστροφές και τη λαιλασία σε μια κανονική οικονομική δραστηριότητα. Το θέμα είναι πώς θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τη βία αυτή, να αφοπλίσουμε τις πολιτοφυλακές, να τις επαναντάξουμε, να μην υπάρχει ατιμορρησία και ταυτόχρονα να υπάρξει συμφιλίωση. Το ερώτημα είναι πολύ δύσκολο. Και τέταρτο ερώτημα πώς ε, οι κατεπίγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες θα καλυφθούν. Και τέλος, ποιος ε, θα είναι ο ρόλος που θα παίξουν ε, οι γειτονικέ χώρες και οι υπόλοιπες χώρες όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, πέραν αυτού που έχει μέχρι τώρα γίνει και είναι ανεπαρκές. Λοιπόν αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα που έχουμε μπροστά μας θα δώσω τον λόγο στον Κούν Φεφάκε, ο οποίος είναι υπεύθυνος του καταπιστεύματος για την Αφρική. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ καταρχάς ε, που αφιερώνετε το χρόνο να συζητήσουμε την κατάσταση στην ε, Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία. από κοινού η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η ΤΕΦΚΟ και αυτό θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Η ΤΕΦΚΟ και η ΕΚΟ. Θα ήθελα να σας θυμίσω ε, Πού βρισκόμαστε. Το 2013 και 2014 η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία αντιμετώπισε τη χειρότερη κρίση που έζησε ποτέ, όπου είχαμε την ε, ε, επαναστατική ομάδα Σέλεκα κατά των ε, στρατευμάτων. Καταρχάς με γαλλικές δυνάμεις, αλλά κατόπιν με δυνάμεις του ΟΗΕ και ειρηνευτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθήσαμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση αυτό δεν αρκούσε και υπήρχε ανάγκη να ακολουθήσουμε και πολιτική οδό. Όσον αφορά την ε, ανάπτυξη θα ήθελα να ε, αναφέρω ε, ότι τον Νοέμβριο του 2016 η Φεντερίκα Μοκερίνη οργάνωσε διάσκεψη όπου η κυβέρνηση παρουσίασε το εθνικό της σχέδιο για αποκατάσταση και ειρήνη. Και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ για, την, τη μετάβαση της κεντροαφρικανικής ε, δημοκρατίας ε, στην ειρήνη. 2015-2016 είχαμε εκλογές χρηματοδοτημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεδομένων των πολύ δύσκολων συνθήκων ε, ήταν πολύ επιτυχής. Και ολοκληρώθηκε έτσι η πολιτική μετάβαση και μπορέσαμε έτσι να αποκαταστήσουμε την ε, τάξη και έχουμε τώρα τον πρόεδρο Ταντέρα και την κυβέρνησή του. Παρά τις εκλογές αυτές, ε, παρά την ε, κινητοποίηση ε, και την μαζική βοήθεια της διεθνούς κοινότητας, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στα τέλη του 2016 αλλά και το πιθανότερο και φέτος είδαμε πολύ σημαντική διάβρωση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια με νέες συγκρούσεις. Ένα στοιχείο εδώ πέρα είναι η ανικανότητα της κυβέρνησης να δώσει καλύτερη ζωή και ασφάλεια στον, στον λαό. Είδαμε λοιπόν και πάλι συγκρούσεις ε, ανάμεσα ε, στις ε, δύο βασικές αυτές ομάδες. Πάνω από 800 άτομα έχουν σκοτωθεί το πρώτο εξάμεινο του 2017. και έχουμε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένων ανθρώπων στην ε, περιοχή. Πρόσφατα εκτοπισμένων. Αυτό ε, αφορά το σύνολο της χώρας εκτός από τον Παγγί. Βλέπουμε συγκρούσεις ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες για ε, πρόσβαση, για έλεγχο και για πρόσβαση σε πόρους, σε διαμάντια, δάση κλπ. Οι συγκρούσεις αυτές λοιπόν συνδέονται με την έλλειψη ε, δημόσιας τάξης και την δυσκολία της ε, κυβέρνησης στο Χαρτούμ να διασφαλίσει αυτά τα βασικά. Έχουμε δει διακοινωτικές και ε, συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές ομάδες συχνά και με ε, θρησκευτικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό, διότι ε, περιλαμβάνει και ε, εκφράσεις μίσους ανάμεσα στις διάφορες ομάδες υπάρχουν κάποιες ομάδες ε, με πολύ, ε, με πολύ συγκεκριμένους αθλητικούς και θρησκευτικούς στόχους και αυτό είναι πολύ ε, ανησυχητικό. Οι δυνάμεις του, του ΟΗΕ κάνουν ό,τι μπορούν για να σταματήσουν τη βία και να προστατεύσουν τους πολίτες, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην, εφαρμογή, στην άσκηση της εντολής της έχουν σκοτωθεί αρκετοί φέτος. Ε, το βασικότερο τμήμα της δύναμης αυτής, της ειρηνευτικής δύναμης Μινούρκα, προέρχεται από την Πορτογαλία. Ελπίζουμε ότι στη Νέα Υόρκη το αποτέλεσμα των συναντήσεων θα είναι ενίσχυση της δύναμης αυτής. Η έκθεση του Προέδρου Κουτιέρης δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα και ελπίζουμε να ακούσουμε περισσότερα από τον συνάδελφό μας στον ΟΗΕ εντός της σημερινής ημέρας. Είναι σαφές ότι ακόμα και με αυξημένο δυναμικό δεν θα μπορέσει η Μινούρκα να διασφαλίσει το σύνολο της περιοχής. Ε, χρειάζεται και μεταρρύθμιση του χρειάζονται σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις και ο ΙΕ θέλει να εκπαιδεύσει ε, δύο με τρεις ταξιαρχίες των εθνικών δυνάμεων. Ήδη έχουμε εκπαιδεύσει δύο, αλλά Ε, θα πρέπει επίσης να γίνει η επανένταξη αυτών των ε, στρατευμάτων στον Εθνικό Στρατό. Ε, θα θέλαμε να επιμηκύνουμε την εντολή κατά δύο χρόνια και να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη για την οικοδόμηση δυναμικού στην αστυνομία σε στενή συνεργασία με τον ΟΗΕ που είναι επικεφαλής σε αυτόν τον τελευταίο τομέα. Η μόνη λύση όμως θα είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση, η ειρήνη με τις ε, ομάδες ε, των ε, επαναστατών και διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Νομίζω ότι είναι κοινή θέση ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ηγηθεί των προσπαθειών αυτών. Έχουμε τώρα μια αξιόπιστη κυβέρνηση που προέκυψε από εκλογές. Χρειάζεται όμως και υποστήριξη από την διεθνή κοινότητα. Και ε, βοηθάμε την κυβέρνηση, έχουμε ε, κινητοποιήσει επιρογνώμονα που θα υποστηρίξει τον Πρόεδρο και ε, που θα ενισχύσει την, την διαπραγματευτική στρατηγική. Έχουμε λοιπόν την πρωτοβουλία της Αφρικανικής Ένωσης να συγκεντρώσει όλες τις γειτονικές χώρες της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας ε, που έχουν πολύ ε, σημαντική ευθύνη στο πλαίσιο αυτό. Η Γκαμπόν, ε, η Κονγκοπραζαβίλ, η Αγγόλα, το Τσάντ και οι περιφερειακές και οι περιφερειακοί οργανισμοί έχουν συγκεντρωθεί. Έχουμε τον οδικό χάρτη της Λιμπρεβίλ, για διαμεσολάβηση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις ένοπλες ομάδες. Είδαμε κάποιες εντάσεις ε, ανάμεσα στην πρωτοβουλία αυτή και το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση και το τι κάνει ο ΟΗΕ. Και γι' αυτό η ε, εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η, εξωτερική, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, την 1η Ιουνίου συγκέντρωσε όλα τα μέρη ώστε να συγκεράσουμε όλες τις πρωτοβουλίες και να υπάρχει συνοχή. Χαιρόμαστε λοιπόν που με τη συνάντηση στις Βρυξέλλες ε, υπάρχει πολύ καλύτερη συνοχή και ότι η διεθνής ε, κοινότητα ε, έχει συσπηρωθεί γύρω από την Αφρικανική Πρωτοβουλία και αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσουν τμήμα αυτής της διαδικασίας. Ποιε είναι λοιπόν οι προκλήσει για τι επόμενε εβδομάδε. Θα πρέπει να φροντίσουμε να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, να ε, έρθουμε σε επαφή με ε, τι ε, με τις διάφορες ενοπλές ομάδες και να εξετάσουμε τα θέματα δικαιοσύνης, ατιμορρησίας και πώς θα βρούμε την ε, σωστή ισορροπία. Αυτό είναι σημαντικό για μας. θέλουμε να υπάρξει δίωξη για τα, για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και υπάρχει αντίθεση απέναντι σε μια γενική αμνηστία αυτό θεωρούμε ότι θα συνεχίσει την βία που έχουμε δει επί τόσο καιρό στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη και συμφιλίωση δεν θα μπορέσει να υπάρξει η ειρήνη. Αυτή είναι η λεπτή ισορροπία που πρέπει να βρούμε όταν εφαρμοστεί η Αφρικανική Πρωτοβουλία μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχει μια Επιτροπή Δικαιοσύνης και Συμφιλίωσης, ε, την οποία στηρίζουμε. Υπάρχει επίσης και ειδικό ποινικό δικαστήριο, σε στενή συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ε, νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν τώρα πια όλα τα στοιχεία και μπορώ επίσης ε, να σας παραπέμψω στην έκθεση του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα αποτελέσει τη βάση για τις έρευνες ε, του Ειδικού Δικαστηρίου, πολύ σύντομα. Συμμετέχουμε ενεργά στις πολιτικές ε, αυτές εργασίες. Βρισκόμαστε καθημερινά σε επαφή με όλες τις ομάδες συμφερόντων στην ομάδα, με τον Πρόεδρο και με τα κράτη-μέλη. Η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι μία από τις περιπτώσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε όλες τις στοιχές πολιτικά, ε, όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, στρατιωτικά κλπ. Ε, είναι μία από τις περιπτώσεις τις ξεχασμένες από τη διεθνή κοινότητα. Φροντίζουμε λοιπόν να μην ε, εξετάζουμε μόνο το κέρας της Αφρικής, τη ζώνη Σαχέλ, αλλά να ασχολούμαστε και με την Κέντρο Δημοκρατία. Εάν ε, πάνε στραβά τα πράγματα εδώ πέρα, θα διαδοθεί η κρίση και σε γειτονικέ χώρε. Γι' αυτό ε, μα ενδιαφέρει και για στρατηγικού λόγου, πέρα δηλαδή από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και αναπτυξιακή βοήθεια, μα ενδιαφέρει να συμμετέχουμε στην προσπάθεια. Θα κλείσω εδώ και είμαι βέβαιο ότι οι συνάδελφοι θα συμπληρώσουν αυτά που είχα εγώ να πω. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω αμέσω το λόγο στην Κάρλα Μοντέση, τη Διευθυντρή, τη Δυτική και Κεντρική Αφρική από την ΓΑΜΑΔΕΛΤΑ Ντεύκο. Δέκα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, θέλουμε να δείξουμε ότι βασιζόμαστε Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι εξελίξεις πολιτικές μπορεί να υπάρξουν, όπως είπε ο Κούν. Δεν θα ασχοληθώ με την ανθρωπιστική κατάσταση, γιατί η συνάδελφος είναι αυτή η οποία έρχεται από εκεί και θα μας παρουσιάσει με λεπτομερή τρόπο την πολύ σοβαρή κατάσταση που υπάρχει στον ανθρωπιστικό τομέα. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου στα θέματα ε, ανάπτυξης και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν για να βγουν από την κρίση. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βασικός υποστηρικτής της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Είμαστε παρόντες και με ανθρωπιστική βοήθεια και με αναπτυξιακή βοήθεια σε όλες τις φάσεις του πολέμου και της κρίσης. Ήμασταν παρόντες επίσης και τη στιγμή εκλογής του νέου Προέδρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εξωτερική Υπηρεσία οργάνωσαν και την διεθνή διάσκεψη για την Κεντροαφρικανική αμέσως μετά ε, την εκκίνηση των προσπαθειών ανοικοδόμησης της χώρας. Συνεργαστήκαμε με τη χώρα, αλλά η ίδια η χώρα δεν είναι σε θέση να δώσει στον εαυτό της ε, την στρατηγική που χρειάζεται. Βέβαια, Έχουμε καθορίσει κάποιες βασικές γραμμές μαζί τους για την ανοικοδόμηση της χώρας, την οποία προετοίμασε η ίδια η χώρα με τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών και εν μέρη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι πιέζουμε τη χώρα να εντοπίσει τις προτεραιότητές της και τις βασικές της στρατηγικές. Είναι σαφές ότι η κατάσταση πέρα από τον ανθρωπιστικό τομέα και η οικονομική κατάσταση είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Έχουμε μια ανάπτυξη πολύ περιορισμένη λόγω ακριβώς της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω την ακαταλληλότητα όλων των ε, υποδομών όπως επίσης και των δομών που απαγορεύουν έτσι όπως είναι σήμερα την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας, ε, τη φορολογία που είναι, τα φορολογικά έσοδα που είναι ανεπαρκή, τον προϋπολογισμό που είναι ανίκανος να χρηματοδοτήσει τα πιο βασικά που χρειάζονται. Συνεπώς λοιπόν η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή σε όλους αυτούς τους τομείς. Πάντως αυτό το πρόγραμμα που έχει προετοιμαστεί υπάρχουν κάποιοι βασικοί άξονες παρέμβασης και σε αυτούς τους βασικούς άξονες η Ευρωπαϊκή Ένωση με ολοκληρωμένο τρόπο από το ανθρωπιστικό κομμάτι στο αναπτυξιακό κομμάτι, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και στην παρέμβαση συνοδείας αν θέλετε και παρακολούθησης των μεταρρυθμίσεων εμείς από τη διάσκεψη και μετά αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε και θα περιοριστώ στα του μέλλοντος και του παρόντος και όχι στα του παρελθόντος. Ήδη υιοθετήσαμε ακριβώς το ΠΙΝ, το Εθνικό Αναπτυξιακό ε, Πρόγραμμα για την απορρόφηση 380 εκατομμύριων. Παρεμβάσεις και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν της ανθρωπιστικής, Πρόκειται για προσπάθειες βελτίωσης της governance, της διακυβέρνησης της χώρας και στον οικονομικό τομέα και στον φορολογικό τομέα. Μια διακυβέρνηση δημοκρατικής φύσης. Πρόκειται επίσης για την υποστήριξη του τομέα της ασφάλειας, της στήριξης της τάξης και της συμφιλίωσης και να διασφαλίσουμε επίσης την γεωργική παραγωγή και να βελτιώσουμε <clears throat> τις συνθήκες εργασίας, να υπάρξει μια ουσιαστική πολιτική δηλαδή παρέμβασης στον τομέα της απασχόλησης, να υπάρξει αποκατάσταση των γεφυριών εκεί που έχουν σπάσει έτσι ώστε να υπάρχει επικοινωνία διάφορα στις, ανάμεσα στις περιοχές της χώρας τον Ιούνιο καταφέραμε επίσης να υποστηρίξουμε, ε, να κάνουμε μια ένεση δημοσιονομική στον προϋπολογισμό, 64 εκατομμύρια, ήδη έχει κατατεθεί το πρώτο τμήμα των 20. Hay un problema con la interpretación en, en inglés. Τα αγγλικά ε, δεν μεταφράζεστε από ό,τι κατάλαβα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με το κανάλι των αγγλικών. Όλα εντάξει. Μπορείτε να συνεχίσετε. Um, Νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να ομιλώ την Ιταλική. Είναι μια ευκαιρία εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές. Λοιπόν, υπήρξε μια πρώτη δημοσιονομική παρέμβαση 64 εκατομμυρίων. Προβλέπεται 20 δόθηκαν ήδη, έτσι ώστε η νέα κυβέρνηση και ο νέος πρόεδρος να καλύψει τις πιο επίγουσες δαπάνες όπως η χρηματοδότηση και η μισθή της δημόσιας διοίκησης και θα ολοκληρώσουμε γενικά τις ε, διαδικασίες ε, για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας, της στήριξης της τάξης και της υποστήριξης των ειρηνευτικών διαδικασιών και των διαδικασιών συμφιλίωσης. Είναι, αν θέλετε, κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία και ε, με τους εκπροσώπους των στρατιωτικών δυνάμεων αλλά και των Ηνωμένων Εθνών και της Μινούσκα έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να βελτιώσουμε αν θέλετε ε, την προοπτική για τις άμεσες ε, ανάγκες στον τομέα των παρεμβάσεων. Τώρα για την άμεση βοήθεια προς τον πληθυσμό της χώρας, όπως ήδη υπόθηκε στην αρχή, να υπογραμμίσω την ύπαρξη του καταπιστεύματος του ειδικού, κάτι το οποίο από το 14 μας επιτρέπει να καλύψουμε κάποιες ε, βασικές ανάγκες. Ε, το καταπίστευμα αυτό θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, θα μεταφέρουμε 45 εκατομμύρια στο Ταμείο Μπικού, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να καλύψουμε τις καταπροτεραιότητες, ε, κατά προτεραιότητα δράσεις, όπως η χρηματοδότηση ή αποκατάσταση των γεφυριών είναι προϋπόθεση για τις περιοχές που είναι απόλυτα απομονωμένες σήμερα, κάτι το οποίο θα επιτρέψει την επιστροφή της δημόσιας διοίκησης εκεί. Επίσης διασφάλιση για την κάλυψη των αναγκών των τροφίμων και βελτίωση του συστήματος υγείας που είναι προβληματικό. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν ε, κάτοικοι της χώρας οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις αυτές. Έχουν ξεκινήσει κάποιες οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες όσο ε, απλές και να είναι βοηθούν τα πράγματα ε, γιατί είχαμε να κάνουμε με πληθυσμούς οι οποίοι είχαν χτυπηθεί άσχημα από στρατιωτικές ομάδες και είχαν διακόψει κάθε οικονομική δραστηριότητα. Στηρίζουμε, όπως είπα, και την κυβέρνηση για να ενισχύσει το θεσμικό της βάρος. Είναι ιδιαίτερα ασθενής η δημόσια διοίκηση και έχει υπάρξει σημαντική βοήθεια και από τα Ηνωμένα Έθνη και από εμά για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και τεχνική βοήθεια συνεργασία με την δημόσια διοίκηση για να πετύχουν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Η πρόκληση σήμερα είναι ότι αυτή η δημόσια διοίκηση να επιστρέψει ουσιαστικά στη χώρα γιατί είναι απούσα σε πολλές περιοχές και να αναλάβει εκ νέου τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των περιοχών αυτών. Αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Σουζάν Μαλεούναβα, προϊσταμένη μονάδα για τη Βόρεια, Δυτική και Κεντρική Αφρική Επιγραμματέλη τα ΕΚΟ και εσείς 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όπως ήδη προείπαν ο Κούν και η Κάρλ, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της Κεντροαφρικανική δημοκρατίας. Επίσης, Είμαστε και ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότε που παρέχουμε ανθρωπιστική συνδρομή, δείχνοντα έμπρακτα την αλληλεγγύη μας προς τον ευάλωτο πληθυσμό τη κεντροαφρικανική δημοκρατία, αλλά και όσου έχουν φύγει σε γειτονικέ χώρες βοηθούμε. Το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε 88 εκατομμύρια για ανθρωπιστική βοήθεια στον πληγέντα πληθυσμό και μόνο φέτος ε, έχουμε ήδη 24 ε, εκατομμύρια για την υποστήριξη ε, στους εσωτερικά εκτοπιστέντες ε, και σε όσους πλήττονται από τις συγκρούσεις εντός κεντροαφρικανικής δημοκρατίας συν την ανθρωπιστική υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους πρόσφυγες που βρίσκονται σε γειτονικέ χώρες και συγκεκριμένα στο Τσάντ και στο Καμερούν. Επομένως, όπως βλέπετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους βασικούς χρηματοδότες ανθρωπιστική βοήθεια στην ανθρωπιστική αυτή κρίση που δυστυχώς ε, είναι ακόμη πολύ οξυμένη. Ε, το 2017 έγινε μια εκτίμηση η οποία έχει αναφερθεί ε, προς τα άνω Μιλάμε για 500 εκατομμύρια δολάρια τα οποία χρειάζονται για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. 30% μόνο ε, έχουμε καλύψει και είμαι βέβαιη ότι και η Νατζάτ ε, που είναι η ειδική εντεταλμένη θα πει περισσότερα. Υπάρχει λοιπόν τρύπα ε, στον προπολογισμό για την στήριξη του πληθυσμού και την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών. Και αυτό είναι άκρο ανησυχητικό, ιδίω στη σημερινή κατάσταση. Ακούσατε πώ έχει κατάσταση πραγματικά έχουμε επιδείνωση και αυτό απαιτεί πραγματικά πολύ περισσότερο τη διεθνή προσοχή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα τη δυνατότητα ε, να βρεθώ ε, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Όλη την εβδομάδα έμεινα εκεί μαζί με διευθυντέ ε, επίγουσων καταστάσεων από τρει οργανισμού. Είδαμε το Hotspot Spria και με την επίσκεψή μα εκεί πραγματικά επιβεβαιώσαμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση. Επιδεινώνεται, οι ανάγκε είναι μεγάλε και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη. Είπε ο Κούν ήδη ότι φέτος Έχουμε πολλά κρούσματα βίας ε, σε διάφορα ε, μέρη, κέντρο, ε, δύση, νότο της χώρας και το Μάιο ιδίως είχαμε πολλές βίες επιθέσεις ε, με αποτέλεσμα αύξηση κατά 50% ε, στον πληθυσμό των εσωτερικών εκτοπιστέντων ατόμων. 600.000 άνθρωποι στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι σήμερα εσωτερικώς εκτοπισμένοι και περίπου 481.000 πρόσφυγες ε, είναι σε γειτονικέ χώρες. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε γυρίσει πάλι στην κατάσταση του 2013 και 2014 είπε και ο πρόεδρος στην αρχή, ότι η κατάσταση αυτή είναι τέτοια όπου ένας στους πέντε κατοίκους της, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας έχει εγκαταλείψει την αιστεία του και καταναγκαστικά εκτοπίστηκε και εξαρτάται από την παροχή βοήθειας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, μια τέτοια κατάσταση σε μια χώρα όπως είναι η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου ο πληθυσμός ήδη είναι πάρα πολύ ευάλωτος για διάφορους λόγους ε, που νομίζω ότι προσπαθούμε εμείς με την αναπτυξιακή μας χρηματοδότηση να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε το εξωτερικό ε, σοκ όπως αυτή η καταναγκαστική εκτόπιση ουσιαστικά σημαίνει ότι ο πληθυσμός αυτός πραγματικά εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ανθρωπιστική βοήθεια. Η εκτίμηση λοιπόν τώρα είναι ότι πάνω από το ίμιση ε, του πληθυσμού της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας απαιτεί διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια. Μιλάμε για 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι εξαρτώνται από την εξωτερική βοήθεια αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην κεντροαφρικανική δημοκρατία μόνο. Όπως είδαμε λοιπόν οι ανάγκες, οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι πραγματικά τεράστιες. Και υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική ανταπόκριση. Η χρηματοδότηση, καλύτερα η έλλειψη χρηματοδότησης, δεν είναι η μόνη πρόκληση. Υπάρχουν πολλές άλλες και μία μείζον πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η πρόσβαση. Πρόσβαση υπό διάφορε έννοιε το εννοώ. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ή αν υπάρχει είναι πάρα πολύ λίγο το δικό δίκτυο. Είναι σε απομακρυσμένε ε, περιοχέ ε, οι εκτοπιστέντε ε, και είναι πολύ δύσκολο να φτάσει κανεί εκεί. Δεν είναι βατή η χώρα αυτή. Πολύ δύσκολη η πρόσβαση λοιπόν. Επίση, λόγω τη αβεβαιότητα και τη ανασφάλεια σχεδόν σε όλη τη χώρα, τα είδαμε και φέτος με τις επιθέσεις στις ανθρωπιστικές οργανώσεις και την, ε, τις εισβολές ε, στα, στις αποθήκες ε, και τη λαϊλασία των χώρων των ανθρωπιστικών οργανώσεων υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση γιατί δεν υπάρχει και επαρκής αποδοχή από τον πληθυσμό των ανθρωπιστικών οργανώσεων, από τις ενόπλες ομάδες, από τη κυβέρνηση. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα με τη δική μας υποστήριξη φέτος. 24 εκατομμύρια σας είπα ήδη έχουν δοθεί ως ανθρωπιστική κατεπίγουσα βοήθεια στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για τον μηχανισμό έγκαιρης αντίδρασης που χρειάστηκε να συγκροτηθεί ώστε να μπορούν οι οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια να φτάσουν γρήγορα στους καταναγκαστικά εκτοπιστέντες που εξαρτώνται ε, για τα βασικά και τα στοιχειώδη αλλά και για παροχή τροφίμων, ε, για τις πρώτες βοήθειες, ε, για την ε, εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης των περιστατικών κτλ. Συνεχίζουμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες που έχουν διαφύγει σε γειτονικέ χώρες, ιδίως στο Καμερούν και στο Τσάντ. Τους δίνουμε βασικά τρόφιμα, δυστυχώς κάτι πολύ αναγκαίο γιατί εξαρτώνται ε, τους παρέχουμε κάποια project για τον τομέα της ασφάλειας και ε, κάποιες δραστηριότητες για να μπορέσουν να έχουν μια πιο υγιή καθημερινότητα και να είναι κάπως πιο αυτάρκης. Τώρα, επειδή η ανθρωπιστική προοπτική ε, είναι ζωφερή για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, θα ήθελα να τονίσω πέντε στοιχεία που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν πραγματικά να βοηθήσουν να, να υπάρξει ε, με μια καλύτερη ανθρωπιστική αντίδραση. Το πρώτο στοιχείο είναι η κατεπίγουσα ανάγκη οι ε, οργανώσεις επιτόπου να μπορέσουν να αναβαθμίσουν τις δυνατότητές τους να παρέχουν γρήγορα ε, μια ανταπόκριση στις ανάγκες όταν αυτές προκύπτουν, ιδίως από μακρισμένες περιοχές, ώστε να μπορούν να αντιδρούν γρήγορα σε αυτές τις αυξανόμενες εκτοπίσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν καταναγκαστικά σε διάφορα τμήματα της χώρας. Το δεύτερο στοιχείο είναι μεγαλύτερος ακόμη συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ε, οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βοήθειας εκεί για να πονηθεί μια κοινή ανάλυση των αναγκών και ένας κοινό σχεδιασμός ανταπόκρισης με σαφείς στρατηγικές προτεραιότητες. Τρίτο στοιχείο σαφής διάκριση μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δράσεων και προσπαθειών, κάτι που θεωρώ must απαραίτητη προϋπόθεση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία και είναι κάτι που σίγουρα θα βοηθήσει να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοχή για, τους διεθνείς, ε, για τις διεθνείς οργανώσεις βοήθειας. Το άλλο στοιχείο είναι να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ αναπτυξιακής ε, βοήθειας και ανθρωπιστικής βοήθειας. Προσπαθεί η Κομισιόν και με το Ταμείο που ανέφερε η Κάλλα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και να υπάρξει καλύτερη ε, ανταπόκριση στις ε, γειτονικέ χώρες, λόγω της παρατεταμένης ε, εκτόπισης, διότι δυστυχώς οι πρόσφυγες που βρίσκονται στις γειτονικέ χώρες δεν φαίνεται να έχουν σαφή πρόθεση άμεσα να επιστρέψουν δεδομένη τη κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η ανθρωπιστική αντίδραση στις γειτονικέ χώρες θα πρέπει να ε, μην είναι μόνο κατεπίγουσα στο χαρακτήρα, αλλά να αναβαθμιστεί και να δούμε τι άλλα μέσα και εργαλεία χρειάζονται για να δώσουμε μια πιο ενδεδειγμένη ε, ανταπόκριση στα προβλήματα, λόγω της παρατεταμένης αυτής κρίσης. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει ε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε διεθνές επίπεδο για την κατάσταση που επικρατεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κατάσταση των προσφύγων ε, στο Τσάτ και στο Καμερούν, προσφύγων από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, είναι μια ξεχασμένη κρίση. Αυτό σημαίνει για εμά ότι χρειάζονται πολύ περισσότερε προσπάθειες ε, για την προβολή, για την ευαισθητοποίηση. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό όμω είναι και πρωτοβουλίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Όπω η σημερινή ενημέρωση εδώ ή το πρόσφατο ψήφισμα που ενέκρινε τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ζητά ουσιαστικά οι διεθνείς ε, χορηγοί να, να δώσουν μεγαλύτερη υποστήριξη για να μπορέσει να ε, δοθεί η απαιτούμενη υποστήριξη σε όλους ε, τους πληγέντες από την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η ώρα για ερωτήσεις ή παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Θα ξεκινήσω εγώ με τη δική μου παρέμβαση και αν θέλει κάποιος άλλος το λόγο μπορεί να το ζητήσει. Για μας λοιπόν η κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι πραγματικά άκρος ανησυχητική. Ε, μόνο ε, αρκούσα να διαβάσω την εκτεταμένη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τις πολλαπλές συγκρούσεις ε, στη χώρα το 2013 και 2014 για να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα πανόραμα μαζικών δολοφονιών. Οι άμαχοι χρησιμοποιούνται ως όπλο πολέμου πέραν της καταστροφικής οικονομικής κατάστασης. Κυρίως όμως βλέπουμε ότι πλήττεται σοβαρά ο αμάχος πληθυσμός. Έχουμε πραγματικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τα οποία διαπράττονται. Δεν έχουν δώσει κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι ειρηνευτικές προσπάθειες. Είχαμε ε, στο Σανεχίδιο τη διαπραγμάτευση μια συμφωνία στον ήλιο και το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικής ε, είχε μια συνάντηση για την κατάσταση εκεί. Τι έχει γίνει ε, η συζήτηση δηλαδή του οδικού χάρτη προχώρησε, ποια είναι η άποψη. Επίσης εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα σταματήσει αυτή η ε, σύγκρουση με την αποστολή περισσότερων στρατευμάτων. Χρειάζεται μια, ένα συντονισμός για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ε, ανάπτυξη, να πάψει ο κύκλος της ατιμορρησίας και να υπάρξει μια επανασυμφίλωση. Το προτείνουν και ε, τα Ηνωμένα Έθνη και ήταν καλή η εξέλιξη σε άλλες περιπτώσεις. Ε, επίσης, οι καταγγελίες σεξουαλικής βίας από τις δυνάμεις διατήρησης της ειρήνης ε, των Ηνωμένων Εθνών. Τι γίνεται με αυτές τις καταγγελίες. Ερευνώνται αυτές οι καταδικαστές αποτρόπες καταγγελίες. Ε, αυτά τα περιστατικά, τα καταδικαστέα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον Φρανκ Έγγελ. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω γαλλικά έτσι για να έχω μεγαλύτερη γλωσσική πολυμορφία. Δύο πράγματα. Το πρώτο για την Αφρικανική Δημοκρατία μιλάμε για πλήρη κατάρρευση του κράτους, των θεσμών και ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό. Και αυτό δεν είναι χθεσινό φαινόμενο, ούτε έχει να κάνει με το Σελέκα και τον, την Μπαλακά και την μεταξύ τους αντιπαράθεση πηγαίνει πολύ πιο πίσω και στις ένδοξες στιγμές, στις παλαιότερες, η χώρα ποτέ δεν είχε περάσει μια φάση πραγματικά διαρθρωτικής ανάπτυξης. Αυτό θα είχε βοηθήσει πολύ. Φυσικά και πρέπει, αν έχουμε πλήρη κατάρρευση, να υπάρξει πλήρη ανασυγκρότηση με τον ένα τον άλλο τρόπο. Μία επανίδρυση, αν θέλετε. Γιατί όπω και να το κάνουμε, το κράτο αυτό δεν υπάρχει ουσιαστικά. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, σκεφτώ εγώ πώ μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον που όχι μόνο δεν μπορεί να βοηθηθεί, αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικά. Και ο ίδιο ο πρόεδρο, ε, όταν ε, πηγαίνει από εδώ και από εκεί, παραπονιέται για την έλλειψη ουσιαστικά ε, των δυνατοτή, της δυνατότητας του να επιβάλλει το οτιδήποτε, χωρίς να υπάρξει θεσμική σύγκρουση, πάρα πολύ δυσεπίλητη, ακόμη και τυπικά, από αυτό το, εμβι... από το κράτος στα σπάργανα. Αλλά ο έλεγχος ουσιαστικά είναι κάτι που δεν τον έχει ο πρόεδρος. Και διαρωτώ με, μήπως χρειάζεται να είμαστε πιο συνεπείς στην υποστήριξη που παρέχουμε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πιστεύετε ότι τα μέσα που διαθέτουμε για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών, των αναπτυξιακών αναγκών που ε, είναι επακόλουθες, ε, για την ασφάλεια αλλά και για την επανίδρυση του κράτους. Αρκούν οι προσπάθειες αυτές. Είπατε ότι δίνονται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι λίγα, αλλά δεν ξέρω, αρκούν. Και είναι αποτελεσματική βοήθεια. Μήπω πρέπει να έχουμε πιο ομαδοποιημένη, συνεπή, συνεκτική προσέγγιση συνεργασία ίσω και με άλλους φορείς που είναι επιτόπου. Αυτή είναι η βασική μου ανησυχία. Και κάτι άλλο. Με εκπλήσει το γεγονός που αναφερθήκατε σε έλλειψη αποδοχής για μια παρουσία υποβοηθητική. Ποτέ δεν είχαμε την εντύπωση ότι δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι εκεί. Θα ήθελα αν έχετε την καλοσύνη να επεκταθείτε λίγο σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε να ακούσουμε και την ειδική εντεταλμένη τη Μινούσκα και θα ήθελα οι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο να μην περβούν τα δύο λεπτά. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Στα αγγλικά θα μιλήσω. Ζητώ συγγνώμη που δεν ε, Παρακολούθησα όλη την συζήτηση, διότι μαζί με την ε, συνάδελφο ήμασταν σε ψηφοφορία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Μας ε, ενδιέφερε όμως ε, το θέμα αυτό, διότι είχαμε, ήταν να συμμετάσχουμε σε μια αποστολή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, η οποία όμως ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Ποια λοιπόν είναι ακριβώς η κατάσταση της διπλωματικής αντιπροσώπευσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παμάκο, και των κρατών μελών. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά, διότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά. Σε πολλές άλλες χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται εντατικά και συχνά μπορεί να κάνει τη διαφορά, για παράδειγμα όπως στην Ιγυρία. Γιατί λοιπόν και ποιο είναι το μάθημα που μπορούμε να μάθουμε, γιατί έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στην κεντροαφρικανική δημοκρατία. Γιατί είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Και ποια είναι τα λάθη από τα οποία μπορούμε να μάθουμε, τι έχει νόημα. Πώς θα μπορέσουμε να δούμε φως στην άκρη του τούνελ. Ευχαριστώ. Muchas gracias, el señor Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είχα πάει πέντε μέρες την προηγούμενη εβδομάδα, έκανα μια αποστολή μόνος μου εγώ. Είπα στους συναδέλφους ότι πρέπει να πάτε κι εσείς. Προφανώς υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας, αλλά είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια επίσκεψη. Ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις τόπου ιδιαίτερα σε σχέση και με τις παρατηρήσεις που έγιναν από τον Λουξεμβούργιο συνάδελφο. Το κράτος δεν υπάρχει κράτος. Αν υπήρξε κάποτε είναι και αυτό. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτό δεν θα το πετύχουμε μόνο με δημοσιονομικές παρεμβάσεις. Βλέπω ότι δίνουμε τόσα στο κράτος όσο και στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες φεύγουν από τη χώρα. Εγώ είμαι υπέρ της αναπτυξιακής, του, του αναπτυξιακή τους ε, ε, ρόλου. Ήμουν πρόεδρος και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνεργασίας για 25 χρόνια, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το κράτος, γιατί δεν υπάρχει. Το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει γραφομηχανές καν, φυσικά δεν έχει υπολογιστές και υπάρχει ένα έγγραφο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τίποτα δηλαδή. Για να αναπτυχθεί λοιπόν το κράτος θα πρέπει εμείς να βοηθήσουμε να υπάρξει κινητοποίηση των υπαλλήλων, να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα πρέπει το Ταμείο Μπίκου να πηγαίνει κατά 70% στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Γιατί θέλουμε φυσικά να ξαναχτίσουμε το κράτος αλλά και την οικονομία. Για το κράτος, βλέπω ότι περνάει η ώρα, απαιτείται στρατός, στρατός της χώρας. Εμείς τους εκπαιδεύσαμε, το κάναμε αποτελεσματικά χάρη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τώρα δεν έχουν εξοπλισμό στη διάθεσή τους και χρειάζονται όπλα φυσικά. Με αυτό το αστείο εμπάργο ε, που υπάρχει και ισχύει για την κεντροαφρικανική δημοκρατία αλλά όχι για τις ένοπλες ομάδες που τις επιτίθενται. Συνεπώς λοιπόν αυτή είναι η προτεραιότητα, προς τα εκεί θα πρέπει να κινηθούμε. Και δεύτερον γνωρίζετε ότι μόνο το 5% αυτού του τεράστιου εδάφους καλλιεργείται. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη της υπαίθρου. Πρέπει να υπάρξει ένα πραγματικό σχέδιο ανάπτυξης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, είναι στα μέτρα μας αν πράγματι το θέλουμε. Να τελειώσω με κάτι. Η Μινούσκα, για θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι, έχει κοστίσει μέχρι τώρα 850 εκατομμύρια. 10.000, 10.000 είναι εκεί. Ενώ με 3.000 τοπικού στρατού που θα έχει υποστηριχθεί από χώρες οι οποίες γνωρίζουν να δώσουν ε, μάχες όπως η ΙΠΑ, η Ρωσία και η Γαλλία θα αποκαταστήσουν απολύτως την τάξη. Ο κύριος Κάλλας, σας ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται να συμφωνούμε όσον αφορά την περιγραφή της κατάστασης ως έχει αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα που τίθεται είναι με τι μέτρα με τι θεσμικά όργανα θα μπορέσουμε να ξαναοικοδομήσουμε το κράτος. Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα, υπάρχει αμηχανία στο θέμα αυτό. Στο παρελθόν ε, ο ΙΕ είχε κάποιες περιοχές τις οποίες διαχειριζόταν προσωρινά μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη. Και η ερώτησή μου είναι, σε συνεννόηση με τον ΟΗΕ, με την Αφρικανική Ένωση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε... Μήπως θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε στα νησιά του Σολομόντα. Πριν 20 χρόνια εκεί είχε καταρρεύσει το κράτος και μέχρι το, φέτος τον Ιούνιο υπήρχε αυτή η περιφερειακή βοήθεια προς, τα, προς τις νήσους Σολομόντα όπου συμμετείχαν η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία. Οι γειτονικέ χώρες συμμετείχαν και επί 15 χρόνια και μέσα σε 15 χρόνια κατάφεραν ε, ε, αυτό το κράτος από το τίποτα να ε, το κάνουν ένα κράτος ε, λειτουργικό. Εάν λοιπόν η Αφρικανική Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι γειτονικέ ε, χώρες συνεργαστούν, μπορέσουν ε, να συνεργαστούν, νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε αποτελέσματα και μαζί με εμπειρογνώμονες, μαζί με τους ανθρώπους από την ανθρωπιστική βοήθεια, να κάνουμε τη δουλειά που δεν μπορούν να κάνουν οι αρμόδιοι στο κράτος αυτό. Θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο, αυτό θα με ενδιαφέρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Καλέρ. Η κυρία Καλέρ, παρακαλώ. Ε, Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν είχα πάρει στη συζήτηση από την αρχή, γιατί ήμουν απασχολημένη σε μια άλλη επιτροπή. Το θέμα όμως της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο γνωρίζω καλά και παρακολουθώ από πολύ κοντά. Είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος, δεν μιλάμε για αυτό τον πόλεμο. Και δυστυχώς υπάρχουν εκατομμύρια θύματα όλα αυτά τα χρόνια, περισσότερα από άλλες συγκρούσεις και σε άλλες περιοχές. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται και σε επίπεδο απώλειας ανθρώπινης ζωής πέρα από την οικονομία, πέρα από την πολιτική, να μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Βλέπουμε ότι το κόστος είναι διαφορετικό για τον καθένα. Η βασική μας προτεραιότητα είναι να σταματήσει η βία, να υπάρξει πραγματικά συμφιλίωση. Τον Ιούλιο του 17 υπεγράφει η συμφωνία του Σαν Ετζίντιο με πάρα πολλές δυσκολίες, όμως άρχισε να τίθεται σε εφαρμογή. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν το εξής. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας. Μπορούμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της συμφωνίας σχετικά με τον αφοπλισμό των στρατιωτικών ομάδων. Και όπως είπαν επίσης οι συνάδελφοι, το κράτος δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε λοιπόν να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα αν δεν υπάρχουν κρατικές δομές θα πρέπει να συνοδεύσουμε τις ε, προσπάθειες για την αποκατάσταση των κρατικών δομών. Πρέπει να βοηθήσουμε τη χώρα να πάει μέχρι τις εκλογές. Και συμφωνούμε και με την προσπάθεια η οποία έγινε μέχρι τώρα να ενισχύσουμε την βοήθεια που δίδουμε για να ενισχυθεί και η δημοκρατία και αυτό θα γίνει μόνο αν αναλάβουν τη μοίρα τους οι ίδιοι οι κεντροαφρικανοί. Σύντομα τώρα περνάμε στις απαντήσεις. Η ειδική εκπρόσωπος, πέντε λεπτά παρακαλώ, γιατί στις 12.30 θα αποχωρήσει η επιμελητία. I will. Uh, um, να απαντήσω σε διάφορες ε, από τις ερωτήσεις. Ε, ο ε, Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Κουτιέρες, ε, θα πάει στο Μπαγκουί την επόμενη εβδομάδα. Είναι λοιπόν σημαντικό το μήνυμα αυτό και όσον αφορά ε, την την ε, βία από πλευράς ε, μελών ε, της, των, της αποστολής του ΟΗΕ και θέλουμε ο, κύριος Κουτιέρες να δώσει τέλος σε αυτή τη συζήτηση. Ε, τέθηκε μια ερώτηση σχετικά με την, παρουσία, με την παρουσία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους λίγους, αν όχι ο μόνος, το μόνο το μόνο θεσμικό όργανο που παρέμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Τώρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης έχει θεσπίσει μια σειρά μέτρων ασφαλείας, τα οποία είναι δαπανηρά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε αυτό, διότι αποφασίζεται και για τον προϋπολογισμό μας. Ήταν όμως σημαντικό να παραμείνουμε και τώρα πια λειτουργούμε κανονικά. Τι να κάνουμε, αυτό ήταν ε, ε, το ερώτημα που ακούστηκε σε όλες τις παρεμβάσεις. Ε, καταρχάς δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε την σημασία των εκλογών. Ναι, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν κρατικές δομές, πραγματοποιήθηκαν όμως εκλογές όπου οι πολίτες έδειξαν ότι ανήκουν σε ένα κράτος και έχουν εκλέξει σε ελεύθερες εκλογές και πολύ πιο ελεύθερα από τις πολλές γειτονικές χώρες ε, Εξέλεξαν λοιπόν τους ηγέτες τους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να οικοδομήσουμε με βάση αυτό. Αυτό αποτελεί δεδομένο. Βέβαια είναι σε πολύ ασθενή θέση ο ε, Πρόεδρος. Υπάρχουν ήδη διάφορες ομαδοποίησεις εντός της κυβέρνησης. Είναι όμως πολύ σημαντικό να ε, στηρίξουμε τον Πρόεδρο. Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο, διότι όλες οι επενδύσεις ε, για ε, να συγκεράσουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες για τις οποίες μίλησα, την Αφρικανική, άλλες χώρες που ήθελαν γενική αμνηστία. Όλα αυτά λοιπόν τώρα με τον οδικό χάρτη της Λιβερβίλ φαίνεται να γνωρίζουμε πού πηγαίνουν. Ε, πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ε, συμφιλίωση, δικαιοσύνη και ατιμορρησία. Τώρα λοιπόν έχουν τεθεί τα σημεία αναφοράς ε, για το πώς θα προχωρήσουμε και βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση και με τον ΟΗΕ και με τις χώρες της περιφέρειας για να φροντίσουμε όλα αυτά να γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, διότι μας πιέζει πολύ ο χρόνος. Κατόπιν έχουμε την υποστήριξη προς ε, την κυβέρνηση. Ε, δεδομένης ε, της ανάγκης να παρουσιάσουμε γρήγορα αποτελέσματα, δεν μπορούμε να βάλουμε όλα τα αυγά μας σε ένα καλάθι, να στηρίξουμε δηλαδή μόνο την κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό να επιτρέψουμε και στον ΟΗΕ να παρουσιάσει γρήγορα αποτελέσματα. Όσον αφορά την ασφάλεια. Η ασφάλεια είναι το σημείο για όλα αυτά. Ε, χρειαζόμαστε ασφάλεια για να μπορούμε να ε, προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Όπως σας είπα, έχουμε την αποστολή ε, κατάρτισης. Ήδη έχουμε καταρτήσει δύο ταξιαρχίες, ε, οι οποίες όμως δεν έχουν κινητοποιηθεί διότι δεν έχουν ε, δύο τάγματα, επειδή δεν έχουν ε, τον απαραίτητο εξοπλισμό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η συζήτηση για το CPSD. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα των όπλων. Υπάρχει εμπάργο όπλων. Έχουν ε, θεσπιστεί όλα τα μέτρα όμως ώστε ο κανονικός στρατός να μπορεί να, ε, να, λάβει, ε, όπλα. Θα κλείσω εδώ διότι μας πιέζει ο χρόνος και είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοι θα προσθέσουν σε αυτά που είπα εγώ. Euh, να συμπληρώσω για το ερώτημα το τι ποσοστό δίνουμε στην κυβέρνηση, τι ε, δίδουμε στις μη κυβερνητικέ. Στα πλαίσια των 310 εκατομμυρίων, τα μισά προορίζονται για την συνεργασία με το κράτος, δηλαδή βοήθεια άμεση και έμεση στην κυβέρνηση, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, να προχωρήσει η ανοικοδόμηση των κρατικών δομών και όπως είπε ο Κούν, δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο βέβαια σε αυτού του είδους τη βοήθεια γιατί η κυβέρνηση όπως είπατε σήμερα δεν έχει και πάρα πολλές δυνατότητες δράσης. Παρεμβαίνουμε λοιπόν με όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας μέσω ακριβώς και του κράτους. Υπογραμμίσατε σωστά ότι οι δυνατότητες του κράτους είναι πολύ περιορισμένες. Συμφωνούμε και γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι πρώτοι δωρητές υπάρχει μια συνεργασία σημαντική για να συνοδεύσουμε και να διασφαλίσουμε τις κρατικές υποδομές και στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Γεωργία και στις συγκοινωνίες γίνεται μια προσπάθεια ανοικοδόμησης και ενίσχυσης των δυνατοτήτων των κρατικών υποδομών έτσι ώστε να επιτρέψουμε στην κρατική εξουσία να ανακτήσει τον έλεγχο του εδάφους του. Γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες είναι εκτός συνθήκων ασφαλείας και κάποιες που είναι και εντελώς ε, μη προσβάσιμες. Συνεπώς λοιπόν ακόμα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, δεν μπορούν να φτάσουν σε κάποιες περιοχές λόγω της έλλειψης υποδομών και λόγω των προβλημάτων ασφαλείας. Επιστροφή του κράτους λοιπόν, ανάκτηση της κρατικής δομής στο σύνολο του εδάφους της χώρας. Και εμείς θα συνοδεύσουμε τη διαδικασία αυτή με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στα εδάφη αυτά και στα πλαίσια της κατά στρατηγικής το κράτος ήταν, είχαμε κατανείμει το κράτος σε τρία διαφορετικά χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο. Τώρα φτιάχνουμε μια νέα ταξινόμηση έτσι ώστε να παρεμβαίνουμε εκεί όπου είναι κατεπίγουσα η ανάγκη παρέμβασης έτσι ώστε να βοηθήσουμε την ανάκαμψη την οικονομική σε συνεργασία βέβαια και με τα θέματα τα οποία έχουν γενικότερα άπτονται της ασφάλειας. Κοιτάξτε στο θέμα της αποδοχής. Είναι σαφές ότι αυτό ανήκει περισσότερο στα ανθρωπιστικά θέματα και δεν είμαι εγώ η πιο κατάλληλη να πω όμως ότι έχουν υπάρξει πάρα πολλές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν προβλήματα αποδοχής από πλευράς του πληθυσμού και των ένοπλων δυνάμεων. Γιατί δεν μπόρεσαν να εξηγήσουν ότι η ανθρωπιστική τους δράση βασίζεται αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές αρχές της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας και όχι σε στρατιωτικές ε, δράσεις, ε, δεν συνδέονται με τη Μινούσκα κτλ. Υπάρχουν κάποιες οργανώσεις οι οποίες έχουν καταφέρει να γίνουν αποδεκτές από τον τοπικό πληθυσμό και έτσι βελτιώνουν την πρόσβασή τους σε αυτόν. Ένα μεγάλο τμήμα δεν το έχουν ακόμα πετύχει. Το θέμα της αποδοχής αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι ότι η κυβέρνηση της Κέντρο Αφρικανικής Δημοκρατίας συζητά ένα νόμο για τις μη κυβερνητικέ που θα περιορίσει πάρα πολύ τα περιθώρια δράσης των διεθνών οργανώσεων και αυτό πάντα έχει σχέση με την αντίληψη που έχουν σε σχέση με τα προβλήματα αυτά. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ατζάτα που είναι ένα και εντεταλμένη του των Εθνών για την πολυδιάστατη ολοκληρωμένη αποστολή θεραπευση για την Αφρικανική Δημοκρατία. Έχετε το λόγο. Merci beaucoup. Euh, l'avantage de parler en dernier, c'est que tout a été dit, euh, donc je vais επειδή έχουν υποθεί τα περισσότερα, εγώ θα εστιάσω μόνο σε κάποια συστήματα τα οποία θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία εντάσσονται στις συλλογικές προσπάθειες που δίνουμε. Κοιτώντας και τους ε, άλλους συναδέλφους, ε, σκεφτόμουν τελικά Ηνωμένα Έθνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε και οι δύο που καθόμαστε εδώ στο τραπέζι, οι δύο οργανισμοί, στην ολοκληρωμένη προσέγγιση. Υπάρχει το triple hat, η τριπλή ιδιότητα μόνο στη, στον ενώ εδώ έχετε περισσότερες ομάδες. Γιατί επιμένω. Σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η αποκατάσταση του κράτους δεν θα λύσει από μόνη τα προβλήματα. Ούτε μόνο αν δούμε τα θέματα της δικαιοσύνης θα λύσουμε όλα τα προβλήματα ή αν είναι επιχειρησιακές από μόνες τους οι συμφωνίες του ΣΕΝ ε, θα λύσουν τα προβλήματα ή μόνο οι στις υποδομές θα λύσουν τα προβλήματα ή και η διάσωση των ζώων από μόνη θα λύσει τα προβλήματα. Διότι σήμερα έχουμε να κάνουμε μια κεντροαφρικανική δημοκρατία που έχει περάσει πολλούς κύκλους βίας και συγκρούσεων. Αυτό έχει περάσει και τον πληθυσμό. Τους χαράκτες πολιτικής, τους φορείς λήψεως αποφάσεων, τους πολιτικούς, τις κοινότητες και τους διάφορους άλλους φόρους που εμπλέκονται. Σήμερα λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Η ανθρωπιστική βοήθεια. Δράτω με πραγματικά τις ευκαιρίες που τις παρουσιάζουμε εδώ για να ευχαριστήσω θερμά την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλληλεγγύη που πάντοτε έδειχνε για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Η γενοδορία των Ευρωπαίων πάντοτε ε, έχει ε, καταδειχθεί απέναντι στους κεντροαφρικανούς για θέματα ανάπτυξης, ασφάλειας, ανθρωπιστικής βοήθειας και πλαισίωσης του πολιτικού διαλόγου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός ε, παράγοντας επιρροής. Θέλουμε να ε, ακολουθούμε δράσεις που θα βοηθήσουν τη χώρα να βγει από την κρίση και οι πολίτες να ζουν καλύτερα. Τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της ε, κρατικής εξουσίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις. Ουσιαστικά μιλάμε για ίδρυση κράτους. Γιατί πράγματι τι να αποκατασταθεί. Δεν υπάρχει κάτι για να αποκατασταθεί. Βέβαια πάντα υπάρχει κάτι να αποκατασταθεί στην Κεντροαφρικανική Και αυτό είναι εμπιστοσύνη όχι μόνο στο κράτος ή στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά στην ίδια τη χώρα και στην ύπαρξη της χώρας και στο μέλλον, στο μέλλον της ότι ως πολίτης ε, της χώρας αυτής έχει σε ένα μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο της προσέγγισης και της προσπάθειας που πρέπει να επιτελέσουμε. Και θα σας εξηγήσω το λόγο. Πρώτον, εμείς, οι πολίτες διαφόρων χωρών, πώς νιώθουμε την παρουσία του κράτους. Δεν αντιλαμβανόμαστε το κράτος ε, με τον ίδιο τρόπο. Σε μια άλλη χώρα μπορεί να σας πούν ότι αν κάποιος με επιτεθεί θα με προστατέψει το κράτος. αν κάποιος μου στερήσει ένα δικαίωμα, θα τον ε, θα προστατέψει ο δικαστής, ο αστυνομικό. Ότι αν είμαι γονέας, ξέρω το παιδί μου μπορεί να πάει στο σχολείο με ασφάλεια. Το κράτος μπορεί να πει επίσης, αν είμαι εγώ ασθενής, μπορώ να πάω στο νοσοκομείο και να έχω μια θεραπευτική αγωγή. Αυτό είναι το κράτος. Δηλαδή στοιχειώδη πράγματα που έχουν να κάνουν όμως και βασικά στοιχειώδη δικαιώματα. Σε δικαιώματα τα οποία όλοι πιστεύουμε. Βασικές υπηρεσίες δηλαδή. Σήμερα, όπως είπε η Κάρλα, έχει γίνει δουλειά πλαισίωσης από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και προσπάθεια ε, υιοθέτηση ρεαλιστικής ε, προσέγγισης. Πραγματικά υπήρξε μεγάλη εφόρια μετά τις εκλογές και σωστά Νομίζω δεν διακεντρεύουμε κάτι να πούμε ή να μην είμαστε πολιτικά ορθοί. Ο το του Αντερά είναι ένας από τους σπάνιους Αφρικανούς πρόεδρους που εξελέγει δημοκρατικά. Άρα έχει νομιμοποίηση δημοκρατική. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα είδος ε, θεσμών ως βάση. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η διάσκευση του ε, Νοεμβρίου 16 στις Βρυξέλλες έβαλε τα θεμέλια για την έξοδο από την κρίση. Ταυτόχρονα όμως οι προσδοκίες δεν βασίστηκαν σε υποθέσεις που σήμερα είναι αληθές, γιατί δεν είναι η σημερινή κεντροαφρικανική δημοκρατία η ίδια με τον Ιούνιο του 2017, όπως μάλλον με τον Νοέμβριο του 2016. Οπόμενος δεν μπορούμε να φανταστούμε ε, πώς μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση ακόμα αυτό, ε, αυτή η βία. Δεν ε, είναι τυχαία. Έχει στρατηγική από πίσω. Γιατί ουσιαστικά δεν θέλει να δοθεί στην ε, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δυνατότητα. Στη δική μας προσπάθεια σχεδιασμού, στη στρατηγική μας και στην ανάλυση μας πρέπει να ε, σωματώσουμε το γεγονός ότι σήμερα πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν συμφέρον να παραμείνει το χάος από ότι είναι αυτοί οι οποίοι είναι σημαντικοί πρωταγωνιστές και εντός και εκτός χώρας που ενδιαφέρονται για να βγει η χώρα από την κρίση. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, από μια μέρα στην άλλη, σε εκθαύματος θα υπάρξει παντού κράτος. Αυτό δεν είναι δυνατόν. Σας το λέω και το εννοώ και αναλαμβάνω και την ευθύνη των λόγων μου. Και ελπίζω να μην ε, με αφήσετε μόνοι μου. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Και επειδή μιλάμε για διάσωση ζώων, ναι, πρώτον, φυσικά και μπορούμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα σημεία που δεν μπορούμε, γιατί υπάρχουν κάποια τμήματα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που τα έχουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους οι ένοπλες δυνάμεις. Πλήρη έλεγχο. Και υπάρχει και ανταγωνισμός τώρα, που δημιουργεί μεγαλύτερη δυναμική, αλλά πολύ αρνητική στην προκειμένη περίπτωση βέβαια. Άρα έχουμε διάφορα κριτήρια. Πού μπορούμε και πού οφείλουμε όταν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δυστυχώ υπάρχουν επιλογές που πρέπει να γίνουν, που είναι δυστυχώς πολλές φορές ε, σε βάρος ε, τη πίστη μα. και υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνών με τη στήριξη των κυβερνήσεων υπήρξε μια πρωτοβουλία για να υπάρχει αυτός ο δικός χάρτης που λέει πράσινη ζώνη. Εκεί είναι η ευτυχία, μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Έχουμε την κίτρινη ζώνη που υπάρχουν πράγματα να γίνουν και κάποιος πρέπει να προσεκτήσει, υπάρχει και η κόκκινη ζώνη. Ναι, όλοι μας οι χορηγοί, οι εταίροι, η διεθνής κοινότητα συμφωνούμε ότι εκεί τώρα όπως έχουν τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και απλά το δεχθούμε με τις επιπτώσεις που έχει αυτό. Και θα σας πω ποιες είναι. Θα είναι ανθρωπιστικές, αλλά αν θέλουμε να τα δούμε ολοκληρωμένα τα πράγματα, όταν υπάρχει μια επίπτωση που άμεσα επηρεάζει μια συνιστόση θα πρέπει να την ενισχύσουμε αυτή τη συνιστόσα από την πλευρά των δυνατοτήτων, της χρηματοδότησης, της παρέμβασης. Αλλιώς, επειδή είναι συγκοινωνούντα τα δοχεία, καήκαμε. Επόμενο, πώς θα ρυθμίσουμε το πρόβλημα της ε, ευάλωτης κατάστασης του πληθυσμού. Η συμφιλίωση δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα γιατί η ειρήνη σταθερότητα δεν θα έρθει απ' έξω. Δεν θα έρθει από το εξωτερικό. Μπορεί να τη σαμποτάρει το εξωτερικό, αλλά όχι να την προκαλέσει το εξωτερικό. Μόνο από μέσα μπορεί να έρθει από όλους τους κεντροαφρικανούς που θα πιστούν, θα κινητοποιηθούν και θα συμφιλειωθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο των προσπαθειών που θα πρέπει να γίνουν. Κυρίε και κύριοι, έχουμε 600.000 εξωτερικούς εκτοπιστέντες και καθένας από αυτούς πολλές φορές έχει εκτοπιστεί. Από το 2013 αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε χανζαπλάστα στην πληγή. Τους βάζουμε σε ένα άλλο στρατόπεδο, τους επιτίθενται, τους πάνε αλλού, τους ξαναεπιτίθενται, τους ξαναπάμε σε τρίτο, τους επιτίθενται. Λοιπόν, πηγαίνουν από το ένα, ε, από τον Άννα στον Καϊάφα. Και Τελικά τι δημιουργείται με όλα αυτά. Δημιουργείται οργή, δημιουργείται αγανάκτηση όταν κάποιο ζει σε τόσο ευάλωτη κατάσταση. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει μίσος που δημιουργείται. Πώ λοιπόν θέλετε να φτάσουμε τελικά στην συμφιλίωση, στην εθνική συμφιλίωση με όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας να βρεθούν βιώσιμες λύσεις για να βγει ο πληθυσμός αυτός από αυτή την ευάλωτη κατάσταση και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς χρηματοδότηση. Η ανθρωπιστική πτυχή ποτέ δεν θα αποτελεί τη λύση. Πρέπει λοιπόν πράγματι εδώ άμεσα να υπάρξει διασύνδεση με το αναπτυξιακό σκέλος και με προτεραιότητες, αλλά και με κάποιες βάσεις, με κάποια θεμέλια. Η βάση της ε, σταθεροποίησης είναι η συμφιλίωση. Για τη δικαιοσύνη μιλήσατε και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Μεταβατική δικαιοσύνη πρέπει να την πλησιώσουμε, να την υποστηρίξουμε. Δεν θα έχουμε από αύριο ε, το δικαστήριο που θα λειτουργεί τέλεια. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει πρόοδος που έχει γίνει, αλλά πρέπει να γίνει κι άλλη η καλύτερη δυνατότητα την οποία έχουμε Νομίζω ότι γνωρίζουμε τις σχέσεις που έχουμε μαζί του. Είναι η καλύτερη δυνατότητα για τη χώρα. Και αν υπάρχει ένας πρόεδρος, έστω και ο μόνος πρόεδρος στην χώρα, ο οποίος πήρε κάποιες ξεκάθαρες θέσεις κατά της γενικής αμνηστίας είναι ο του Αδέρα. Γιατί σήμερα αν η ατιμορρησία κυριαρχεί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αφοπλίσουμε. Γιατί το να παίρνει κανείς μία χατζάρα ή μία καραμίνα μόνο και μόνο για να εκδικηθεί και αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Πρέπει λοιπόν αντίθετα να προχωρήσουμε προς μία παραδοσιακού τύπου θεσμική μορφή δικαιοσύνης. Τώρα για τα θέματα ασφαλείας. Φυσικά υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μουνίσκα. Όλες οι πλευρές συμμετέχουν και έχει υπάρξει πρόοδος γιατί το Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Άμυνα ενεκρίθη, υπεγράφει. Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι πλέον και ταυτόχρονα η ενίσχυση των δυνατοτήτων της αστυνομίας και της ανάπτυξης των εσωτερικών δυνάμεων ασφαλείας προσαρμόστηκε. Μια διαφωνία που έχουμε είναι ότι αυτή στιγμή έχουν πάρει τις θέσεις τους οι να υπάρξουν 20 αστυνομικοί και 20 χωροφύλακες, γιατί η Μινούσκα δεν μπορεί να είναι παντού και δεν οφείλει να είναι παντού. Μηδενική ανοχή λοιπόν. Να θυμίσω όμως εδώ τρία πράγματα. Πρώτον, δυστυχώς, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο εσωτερικό και των ειρηνευτικών δυνάμεων, αλλά και στο εσωτερικό των μη κυβερνητικών. Πρέπει να καταγγείλουμε όλες τις περιπτώσεις χωρίς διακρίσεις, και οι δράσεις να αφορούν όλο τον κόσμο. Σε σχέση με τις δράσεις αυτές ε, πρέπει να δημιουργηθεί μια διοικητική μονάδα έρευνας έτσι ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες αποφάσεις. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, σας συγκετεύω. Αυτό δεν θα πρέπει να σας κάνει να ξεχνάτε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις είναι αυτοί που προστατεύουν τους πολίτες σήμερα ότι οι, αυτοί είναι που αποτρέπουν τις φαγές, ότι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν με τη δική τους ζωή την υπεράσπιση των διαδικασιών σταθεροποίησης της κεντροαφρικανικής δημοκρατίας. Ας μιλήσουμε για το ΕΣΥΑ λοιπόν, αλλά να μην ξεχνάμε αυτά τα οποία κάνει η πλειοψηφία ε, των ειρηνευτικών δυνάμεων, να προστατεύσει την ειρήνη και να δώσει μια ευκαιρία ακριβώς για την αποκατάστασή της. Ευχαριστώ την ειδική εκπρόσωπο της Μινούσκα. Ευχαριστώ λοιπόν και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την εκπρόσωπο της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Σχέσεων γιατί αναφερθήκαμε σε ένα θέμα το οποίο δεν μας απασχολεί ιδιαίτερα και προσπαθούμε να βρούμε τι λύσεις μπορεί να υπάρξουν θα συναντηθούμε στο Στρασβούργο στις 23 Οκτωβρίου.